Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Δεν είμαι η κυρία Γκρέσλε, είμαι ο Μάρκος Πίπερ και δεν φαντάστηκα ότι δεν θα ερχόταν η κυρία Γκρέσλε, αλλά δεν ήρθε. Η κυρία Γκρέσλε, και συνεχίζω στα γερμανικά, ασθενή. Έχει σοβαρή γρήπη. Περαστικά της, της ευχόμεθα όλοι και θα προσπαθήσω να την αντικαταστήσω επαξίως. Είμαι υπεύθυνο ε, και για την κατάρτιση της έκθεσης για την χρηματοδότηση των ΜΚΟ για το Κοινοβούλιο. Οπότε συνδυάζω δύο ιδιότητες σήμερα το απόγευμα ε, χωρίς την κυρία Γκρέσλε δυσκολεύομαι λίγο, αλλά ε, ίσως ε, έχει κάποιο νόημα να το αναλάβω εγώ. Χαίρομαι για το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται μέσω της παρουσίας σας εδώ. Είναι πολύ άριθμοι συνάδελφοι. Να εξηγήσω λίγο ε, το ιστορικό του θέματος και γιατί μας απασχολεί. Η έκθεση ελέγχου προϋπολογισμών είναι φύση υπεύθυνη για την διαφάνεια της χρυσής των ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε πολλά προγράμματα Έχουμε κάνει ρυθμίσεις πολύ διαφανείς στα διαρθρωτικά ταμεία. Για παράδειγμα, υπάρχει η διαφάνεια του τελικού ωφελουμένου κάθε ε, ε θα πρέπει να δημοσιεύεται στο διαδίκτυο όταν λαμβάνει διαρθρωτικά ε, κονδύλια. Μας ενδιαφέρει να γίνεται αυτό στα κράτη-μέλη. Και όταν ε, γίνεται η διαδικασία απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάντοτε δημιουργούνται προβλήματα με τα κονδύλια στη Γεωργία, ε, τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων. Τώρα όμως, τα τελευταία χρόνια, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Αυτό που είναι λιγότερα εγκόγνητα ακόμα, σχετικά, είναι η χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανώσεων και η, η χνηλασιμότητα, αν θέλετε, των κονδυλίων και της τύχης τους. Έχουμε την εντύπωση ότι κάθε γενική διεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει αυτό που νομίζει εκείνη σωστό η κάθε μία κάτι διαφορετικά. Ε, δεν θέλουμε βεβαίως ε, να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις εδώ, αλλά ούτε κατηγορούμε κανέναν, αλλά διαδικαστικά δεν ε, είναι ίδιες οι διαδικασίες σε ό,τι αφορά την, την την διαφάνεια ε, στον τομέα αυτό. Ιδιαίτερα ε, το έχουμε εμεί αυτό το πρόβλημα γιατί είμαστε υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των κονδυλίων. Ένας λόγος λοιπόν που αποφασίσαμε να ασχοληθούμε είναι αυτός. Δεύτερος λόγος. Ανησυχούμε σε σχέση με την υποστήριξη των ΜΚΟ και σε ποιο βαθμό προχωρεί αυτή. Ε, Εμεί ε, έχουμε στην Ευρώπη διάκριση των εξουσιών όπου η Κομισιόν είναι η εκτελεστική εξουσία και το Κοινοβούλιο η νομοθετική. Ε, πώς γίνεται λοιπόν η εκτελεστική εξουσία να διαθέτει κονδύλια, να διαθέτει τεχνογνωσία ε, και να επηρεάζει την νομοθετική εξουσία. Σε πολλές χώρες, σε πολλές υπήρους δεν συνηθίζεται αυτό. Στην Ευρώπη επιτρέπεται αλλά πολλές φορές με το σύστημα αυτό χρειάζονται πληροφορίες για να κινηθούμε μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος, ιδιαίτερα όταν αναμένεται από εμάς ως θεσμικό όργανο να επιχειρηματολογούμε αντικειμενικά τεκμηριωμένα. Και γι' αυτό για αυτούς τους λόγους πρέπει να θέτουμε και πολλά ερωτήματα. Χαίρομαι πάρα πολύ διότι έχουμε σήμερα πολλούς εξέχοντες ε, καλεσμένους και θα ήθελα να τους δώσω το λόγο και πρώτα απ' όλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία, ελπίζω να το η κυρία Βικτόρια Ζήλ Κασάντο είναι ε, η πρώτη ομιλήτρια. Χαίρομαι που ήρθατε και από την ε, πλευρά της Κομισιόν θα μας πείτε πώς υποστηρίζονται από εσάς οι ΜΚΟ, τι διαδικασίες ακολουθούνται και τηρούνται και πώς ρυθμίζονται τα θέματα μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Πρώτη δήλωση λοιπόν, πρώτο εισαγωγή θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα ακούσουμε τους υπόλοιπους ομιλητές, ε, θα ακολουθήσει συζήτηση με ερωτήσεις και θα δούμε και την προοπτική άλλων ε, θεσμικών οργάνων, το ελεγκτικό συνέδριο και θα δώσουμε το λόγο και σε εκπροσώπους των ΜΚΟ. Ε, προσβλέπω σε ενδιαφέρουσα ακρόαση και δίνω αμέσως το λόγο στην Τζιλ Κασάδο. Για 10 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να έρθω εδώ, να συζητήσω μαζί σας ε, επί μιας εξαιρετικής εκθέσεως ε, την οποία έχετε εκπονήσει. Είχαμε τη δυνατότητα και ε, τον προηγούμενο μήνα να συζητήσουμε με τους συμβούλους τους οποίους είχατε ορίσει και να σας δώσουμε πληροφορίες βάσει των επιθυμιών σας. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ ε, επί του τι κάνουμε αυτή τη στιγμή σε σχέση με την χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, κάποια στοιχεία δηλαδή ε, χρηματοδότησης, αλλά και κάποια στοιχεία που αφορούν την εκτινασιμότητα και την διαφάνεια. Ε, δεν θα πω, δεν θα έτσι, αναφερθώ αναλυτικά σε αριθμητικά στοιχεία. Θα ήθελα περισσότερο να σας παρουσιάσω τι έχουμε προτείνει ε, ως περιεχόμενο της νέας προτάσεως ε, χρηματοδότησης. Ε, έχουμε ξεκινήσει ήδη την διαπραγμάτευση και με το Συμβούλιο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, οι πρώτες, ε, ε, οι πρώτες θέσεις είναι θετικές. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις πρώτες διαπραγματεύσεις, τις άτυπες και θα προχωρήσουμε και στις επίσημες διαπραγματεύσεις και βεβαίως θα θέλαμε έγκαιρα να μας υποβάλλετε τις προτάσεις σας. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Νομίζω ότι και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο Συμβούλιο, ίσως λιγότερο το Συμβούλιο, ε, θεωρούν ότι το, ο ρόλος που μπορούν και πρέπει να παίξουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι σημαντικός. Όχι μονάχα μας βοηθούν στην ε, υλοποίηση των πολιτικών μας, αλλά αποτελούν και ένα πάρα πολύ καλό think tank ε, που μας βοηθά στο έργο ανάπτυξης πολιτικών. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις συμμετέχουν λοιπόν ε, στη διαδικασία υλοποίησης και εφαρμογής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και εξ αυτού ο, ο ρόλος τους είναι σημαντικό εντός των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε αναπτύξει και διάφορα, διάφορους τρόπους και εργαλεία συνεργασίας. Πρέπει να πούμε ότι αυτές οι διάφορες ε, μέθοδοι ε, αφορούν ε, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που τις χρησιμοποιούν βεβαίω. Μιλάμε για οργανώσεις με τις οποίες έχουμε συνεργαστεί επί έχουμε αναπτύξει αυτό που ε, ονομάζουμε εμείς ε, ε, συμφωνία πλαίσιο εταιρικής σχέσης, framework partnership agreements, που ακριβώς ε, ε, ε, αντιπροσωπεύει και την εμπιστοσύνη που έχουν οι δύο πλευρές, η μία προς την άλλη, κυρίως σε τομείς όπως είναι η ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά μερικές φορές και όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Σημαντικό είναι να πούμε ότι όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις προς τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι δημόσια διαθέσιμες, δηλαδή διέπονται από το σύστημα ζήτημα ε, δημοσιονομικής ε, διαφάνειας ε, δημοσιοποιούμε τα χρήματα, τα οποία τους πόρους, οποίους, τα, τα κονδύλια τα οποία δίνουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ε, γίνει ε, σαφές ότι αυτό το σύστημα δημοσιονομικής ε, διαφάνειας προήλθε και από την προσπάθεια του Κοινοβουλίου ήδη από το 2010 ε, και, τώρα αλλά και στο μέλλον ε, θα εξακολουθήσουμε να βελτιώνουμε τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε πληροφορίες και δημοσιοποιούμε τις πληροφορίες ε, μέσω αυτού του συστήματος δημοσιονομικής διαφάνειας, το FTS. Να σας δώσω κάποια στοιχεία σχετικά με τις περσινές χρηματοδοτήσεις να σας πω ότι δεν δίνουμε πληροφορίες σχετικά με κονδύλια τα οποία ε, δίνονται υπό το κεφάλαιο 1α ε, που είναι ε, κυρίως προγράμματα του ορίζοντα 2020, Εράσμους κλπ. Έχετε όμως εδώ στη διαφάνεια που σας δίνω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει ορισμός ενωσιακός ε, σε σχέση με τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ε, δεν υφίσταται αυτό, γιατί τα συστήματα στις εθνικές νομοθεσίες, δηλαδή, διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους, οπότε η Κομισιόν απεφάνθη ότι είναι περίπου αδύνατον να παράσχει τέτοιου είδους συνολικό ορισμό που και βασιζόμαστε στον ορισμό που δίνει το Κοινοβούλιο. Οι πληροφορίες που δίνει η Κομισιόν για τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις ε, βασίζονται αφενός ε, εις τις δηλώσεις τις οποίες οι ίδιες οι οντότητες υποβάλλουν ως μη κυβερνητικέ οργανώσεις αυτό που ελέγχουμε είναι ότι πρόκειται για ε, ε, ιδιωτικού δικαίου οργανώσεις, ε, οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου και ότι πρόκειται επίσης για οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτό το ελέγχουμε και εμείς. Το κύριο μήνυμα αυτής της διαφάνειας είναι ότι μιλάμε για 1,2 δις, εκ των οποίων το 50% περίπου ε, έχει δοθεί στις ε, ε, πρώτες 50, top 50, στην ομάδα των 50. Υπάρχουν όμως και άλλες οργανώσεις με τις οποίες έχουμε 1.500 συμφωνίες και θα δείτε περίπου το, το μεγαλύτερο ποσοστό μάλλον έχει δοθεί ε, στο, στην επικεφαλίδα 4 Global Europe. Τώρα, όσον αφορά τα προγράμματα, τα οποία κατά προτεραιότητα ε, στα οποία κατά προτεραιότητα μας βοηθούν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ε, εκεί θα βρείτε ε, την ανθρωπιστική βοήθεια, την αναπτυξιακή βοήθεια και βεβαίως και τα εργαλεία για την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπετε εδώ στη διαφάνεια ότι παραπάνω από το μισό του κύκλου είναι, αντιπροσωπεύει την ανθρωπιστική βοήθεια και μετά όλα τα υπόλοιπα. Είναι πάντως γεγονός ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις υποστηρίζουν ε, και την ε, Κομισιόν στην ανάπτυξη νέων πολιτικών. Ε, στην επόμενη τώρα διαφάνεια, που είναι και η τελική με, με αριθμητικά στοιχεία, ε, βλέπετε και τον τρόπο με τον οποίο έχει προχωρήσει ε, η χρηματοδότηση. Ε, δηλαδή όχι ακριβώς το πόσα δίνουμε, αλλά τον τρόπο με τον οποίο τα δίνουμε. Εδώ θα διαπιστώσετε ότι 96 και κάτι της 100 δίνονται εν είδη δανείου, grant επί συγκεκριμένων προγραμμάτων δράσης, δηλαδή ε, χρηματοδότηση ενίδη δανείου για συγκεκριμένη δράση επιτόπου που θα ε, υλοποιηθεί από τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις ε, δίνουμε και κάποια μη επιχειρησιακά δάνεια, έτσι ώστε να κρατήσουμε ζωντανές κάποιες οργανώσεις και με 2, κάτι τα δίνουμε έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν συμβόλαια αλλά διαπιστώνεται ότι εδώ έχουμε στο κάτω μέρος της διαφάνειας και τις ε, κορυφαίες τρεις μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες έχουν ε, χρηματοδοτηθεί και το έτος 2015. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία τα γνωρίζετε ήδη, σας τα έχουμε κοινοποιήσει ήδη και τον προηγούμενο μήνα, ε, αλλά τώρα βρίσκονται πλέον και στην δημοσιοποιημένη μορφή της έκθεσης και στο μέλλον θα σας παρουσιάσουμε ε, και τα όσα προτείνουμε στους ε, συνομοθέτες ε, για το μέλλον όσον αφορά την συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην υλοποίηση των νοσιακών πολιτικών αφενός και αφετέρου όσον αφορά την απλούστευση των διαδικασιών προτείνουμε μέτρα ε, σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας υλοποίησης. Ε, προτείνουμε κάποιες ε, δράσεις απλούστευσης στην πρώτη φάση της υποβολής δηλαδή της αίτησης. Ας πούμε εδώ προτείνουμε να περιοριστούν οι απαιτήσει κάποιων χρηματοδοτικών ε, και διοικητικών ε, εντύπων από τη στιγμή που ενδεχομένως ε, μπορεί να υπάρχουν ήδη βάσει εθνική νομοθεσία. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να μην ζητούμε ξανά τα έγγραφα τα οποία έχουν ήδη, βρίσκονται ήδη στην αρχική τους αίτηση. Επίσης θα πρέπει να αναγνωριστεί η εργασία εργασία των εθελοντών. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν πρόσβαση σε κονδύλια ε, και επομένως βασίζονται στην εργασία των εθελοντών. Αναπτύξαμε λοιπόν και ένα άρθρο έτσι ώστε ε, κάποια κόστη να μπορούν πλέον να είναι επιλέξιμα Επίσης, να σας πω ότι όχι μονάχα δουλεύουν για μας ε, ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, εργάζονται ταυτόχρονα ε, και για άλλους διεθνείς οργανισμούς, ενδεχομένως και για εθνική για την εθνική ε, ε, διοίκηση ε, και επομένως εμείς θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να περιορίσουμε τα διάφορα επίπεδα ελέγχου που είναι πολλαπλά έτσι ώστε να γίνεται καλύτερα η αξιολόγηση και να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι απαιτήσει υποβολής αιτήσεων, συγγνώμη, εκθέσεων και παρακολούθησης σε μερικέ ε, περιπτώσει, πρέπει να σα πω ότι οι μη κυβερνητικές ε, ε, διαπανούν περισσότερο χρόνο ε, για να αντιμετωπίσουν του διάφορου οικονομικού ελέγχου και του διάφορου παντό είδου ελέγχου που πρέπει να αντιμετωπίσουν παρά για να κάνουν τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνουν. Δηλαδή μερικέ φορέ δύο και τρει φορέ πρέπει να κάνουν να υποβάλουν την ίδια έκθεση με λίγο διαφορετικό τρόπο. Εδώ θα δούμε πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή. Επίσης, στο μέλλον θα προσπαθήσουμε σταδιακά ε, να περάσουμε στα e-grants, ε, και δηλαδή η ηλεκτρονική διαδικασία για τα δάνεια και για τις ε, αναθέσεις. έτσι ώστε Ε, έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει και η νομική ε, ε, δυνατότητα αλλά και η οικονομική και η λοιπή ικανότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να τα αποθηκεύουμε στο ίδιο σημείο έτσι ώστε να μην γίνονται διπλή και τριπλή έλεγχη για το ίδιο πράγμα. Επίσης, μετά το 2020 ε, θα ξεκινήσει μια ακόμα πιο καλά οργανωμένη ε, εργασία γιατί θα υπάρχει εναρμόνιση διαφόρων διαδικασιών, ανθρωπιστικής βοήθειας κλπ. Και ούτως ή άλλως ε, δεν χρειάζεται κάθε φορά να αλλάζουν ε, τα πράγματα. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, ξέρουν ε, πώ να αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις και δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε του ελέγχους. Αυτά γενικά. Σα σας έδειξα κάποια αριθμητικά στοιχεία. Σας είπα ποια τροχιά θέλουμε να ακολουθήσουμε και στο μέλλον και ελπίζω να συνεχίσουμε και την καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εισαγωγή από την κυρία Ζήλ Κασάδο και προχωρούμε τώρα στους συμβούλους που ετοίμασαν μελέτη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Προκαταρκτικά να κάνω μια ερώτηση. Α, ποιος η κυρία, ο κύριο Άκερμαν ή η κυρία Περό θα κάνουν την παρουσίαση. Πού, είστε, πού κάθεστε και δεν σας βλέπω. Ε, ποιος θα κάνει την παρουσίαση, ο κύριος Άκερμαν ή και οι δύο. Ο κύριος Άκερμαν. Να σας κάνω λοιπόν μια ερώτηση καταρχήν. Η Κομισιόν δεν απάντησε δυστυχώς το αρχικό μου ερώτημα. δηλαδή σε ποιο βαθμό τα κονδύλια που αναφέρθηκαν και είναι εντυπωσιακά και που πηγαίνουν στις μεγάλες ΜΚΟ, πώς διοχετεύονται μετά με τη σειρά τους σε μικρότερες ΜΚΟ. με ένα σύστημα παρακολούθησης. Γιατί για τις μεγάλες ξέρουμε, αλλά ορισμένες μικρές νιώθουν μειονεκτικά σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που λαμβάνουν. Τι γίνεται στο δεύτερο βήμα, όταν έχουν λάβει οι ΜΚΟ οι μεγάλες τα κονδύλια, πώς μετά τα διοχετεύουν, πώς κατανέμονται στις μικρότερες ΜΚΟ. Υπάρχει τεκμηρίωση και διαφάνεια και για τη διαδικασία αυτή. Αυτή είναι μια ερώτηση που ήθελα να θέσω ευθύ εξ αρχής. Έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε τη μελέτη. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω στην ερώτησή σας πρώτα για την έκθεση που έχουμε δημοσιεύσει. Από τη σελίδα 18 με 20 ασχολούνται με τα θέματα της διαφάνειας στον τομέα των χρηματοδοτικών και περιλαμβάνονται ορισμένοι περιορισμοί Καλό είναι να μπορεί κανείς να συμβουλεύεται αυτή την βάση δεδομένων, αλλά όταν ξεκινάει να τα αναλύει σε επίπεδο λεπτομέρειας, αντιμετωπίζει εμπόδια, τα οποία του το απαγορεύουν ουσιαστικά. Δεν είμαι λοιπόν βέβαιος από την παρουσίαση η οποία έγινε, αν πράγματι προβλέπονται κάποια βήματα για να επιληθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πάρα πολύ συχνά η κατανομή των χρηματοδοτήσεων από τα κέντρα συντονισμού ε, στους εταίρους του κονσόρτιουμ δεν είναι ε, σαφής. Ίσως να μου διέφυγε κάτι. Είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσετε λοιπόν στο άμεσο μέλλον, καλό θα ήταν. Ε, κατανοώ ότι το θέμα είναι περίπλοκο βέβαια. Είναι ένα θέμα το οποίο εμπεριέχει επιμέρους περίπλοκες ρυθμίσεις και δεν αντιμετωπίζεται με πολύ εύκολο τρόπο. Um, yes, so this, short uh, Μια σύντομη παρουσίαση λοιπόν για τα δύο θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόταση προγράμματος. Ο τίτλος της μελέτης είναι «Δημοκρατικός έλεγχος και δημοσιονομικός έλεγχος των ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό». Έχει σημασία να πούμε ότι δεν πρόκειται για έναν λογιστικό έλεγχο. Α, οι πληροφορίες τις οποίες λάβαμε μας δείχνουν ότι έγινε δυστυχώς κατανοητή η προσπάθειά μας σαν προσπάθεια ελέγχου και εποπτείας και επίσης τέθηκαν και θέματα συμμόρφωσης προς συγκεκριμένες γραμμές τήρησης ορισμένων γραμμών, ενώ δεν ήταν αυτός ο στόχος. Απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να πω ότι τα βασικά σημεία της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχουν πάρα πολύ περίπλοκες ε, και διευρυμένες διαδικασίες ελέγχου, εποπτείας ε, και περιγραφής ε, των μορφών χρηματοδότησης. Και υπάρχουν και συστήματα άμεσης εξαίρεσης και διακοπής. Υπάρχει όμως μια πολλαπλή τυπολογία η οποία χρησιμοποιείται Σαν παράδειγμα στα πλαίσια του ε, Financial Transparency System είναι πολύ δύσκολο με τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε να κάνουμε μια συγκεκριμένη ανάλυση των πολιτικών που ακολουθούνται. Υπάρχουν αρκετές διαφορές μάλιστα και αντιθέσεις ανάμεσα στο σύστημα το ίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι πολύ ε, δύσκολο να μπορέσει κανείς να συσχετίσει τις πληροφορίες τις οποίες παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σαν παράδειγμα η αναδιανομή των δανειοδοτήσεων δεν καταγράφεται. Μερικές φορές μπορεί να βρει κανεί στοιχεία, αλλά δυστυχώς είναι ένας γενικός αριθμός, χονδρικός αριθμός, ο οποίος δεν δείχνει την επιμέρους κατανομή. Αντιμετωπίσαμε επίσης και μία περίπτωση όπου ίσως να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες των κανόνων ανάμεσα στις διαφορετικές υπηρεσίες της Επιτροπής. Και επίσης ένα θέμα το οποίο κάνει δύσκολη τη ζωή των ΜΚΟ είναι η έλλειψη διαφάνειας και η έλλειψη σεβασμού των κανόνων. Κάτι το οποίο καθιστά πάρα πολύ δύσκολο το να σεβαστεί κανείς τους συγκεκριμένους κανόνες. Για τα θέματα της αναδιανομής ε, το σύστημα διαφάνειας θα έλεγε, εκπροσωπείται με το σημεάκι στο αριστερό τμήμα της ε, διαφάνειας. Στην ουσία χρηματοδοτείται ένας ε, συντονιστικός οργανισμός, μια μικιό συντονιστική. Είναι ένα μαύρο κουτί βέβαια, όταν πηγαίνει κανείς στις ιστοσελίδες των επιμέρους συντονιστικών μικιών και ζητάει να μάθει πώς διανέμονται τα χρήματα, ε, βλέπει ε, περιγραφές δραστηριοτήτων, βλέπει περιγραφές συγκεκριμένων δράσεων, αλλά είναι πολύ δύσκολο να αθροίσει όλα αυτά τα στοιχεία μαζί. Βρήκαμε λοιπόν ε, ότι υπάρχει μια περιπλοκότητα στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν και χρηματοδοτούν, τροφοδοτούν τα δίκτυα οι συντονιστικές μικιο. Υπάρχουν ε, πολλές φορές σχέσεις ανάμεσα στους εταίρους, του συμβαλωμένους, οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρες και έπρεπε πολλές φορές όταν κάποιος ήθελε στοιχεία να τα ζητάει ξεχωριστά. Τώρα, σε σχέση με το ποιος κάνει τι με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, είναι πολλές φορές δύσκολο να βρει κανείς τη σωστή ενημέρωση. Ταυτόχρονα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να συλλέξει τις πληροφορίες από τα FTS από τις διαφορετικές υπηρεσίες της Κομισιόν και από τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας των ΜΚΟ. Υπάρχει εδώ μια σαφής έλλειψη διαφάνειας. Εδώ συνδέεται φυσικά η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεμονωμένες ΜΚΟ, αλλά πολλές φορές είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τη σχέση αυτή, τη σύνδεση αυτή. Η ΜΚΟ δίνουν διαφορετικά επίπεδα θα έλεγα της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ιστοσελίδες τους. Πολλές ΜΚΟ βάζουν πάρα πολύ μικρά σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι δύσκολο να τα δει κανείς. Λοιπόν, η αξιολόγηση των πληροφοριών λοιπόν ήταν σχετικά περιορισμένη όταν ήταν διαθέσιμη για τη λεγόμενη e-visibility. Ε, εδώ είναι ένας τομέας στον οποίο κανονικά ε, βλέπει κανείς ε, αν οι ΜΚΟ συμμορφώνονται με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Η αλήθεια είναι ότι πολλές ΜΚΟ παίρνουν πάρα πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένες από αυτές, και εκεί υπάρχει ένα πιο σαφές επίπεδο επιθυμητό, αν θέλετε, ορατότητα σε εισαγωγικά της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Οι κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν για την ορατότητα, την δημοσιοποίηση, του, στο σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενισχυθεί. Σχετικά με τις συστάσεις τώρα, εμείς αναγνωρίζουμε ότι πράγματι το να καταλήξει κανείς σε μια συμπεφωνημένη μορφή ορισμού των ΜΚΟ ή των προτέρων είναι κάτι το δύσκολο. Το να μπορέσει επίσης να αναλύσει κάποιος την χρηματοδότηση ίσως θα πρέπει να κάνει το βήμα της κατάληξης σε ορισμένες συμφωνίες, τουλάχιστον για τις διαφορετικές μορφές των οργανισμών αυτών, χωρίς να μιλήσουμε υποχρεωτικά για ΜΚΟ και να υπογραμμίσουμε τις οργανώσεις οι οποίες δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για περαιτέρω ανάλυση, όπως σαν παράδειγμα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά Ινστιτούτα, κάτι το οποίο έκανε και η συγκεκριμένη έρευνα. Ένα ενιαίο συγκεντρωτικό αν θέλετε σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταγραφή και τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων είναι κάτι το οποίο ε, θα ήταν πιο εύκολο να κατανοηθεί. Αλλά όπως σας είπα η προσπάθεια αυτή προφανώς είναι μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Σε μία περίπτωση κατά τη διάρκεια της μελέτης είδαμε ότι το feedback το οποίο είχαμε μας έδειξε ότι αντί να εξαρτώμεθα από τα στοιχεία που δίδουν κάποιες οργανώσεις, τουλάχιστον για τις μεγάλες οργανώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πιο προληπτικό τρόπο θα πρέπει να ε, εποπτεύει την κατάσταση, αλλά αναφέρομαι κυρίως στις, ε, ε, στους οργανισμούς που παίρνουν μεγάλες χρηματοδοτήσεις. Και τέλος να ξαναμιλήσω για την εικόνα της Ένωσης, την ορατότητα της Ένωσης, δεν είναι μόνο το σήμα, αλλά να ε, ενημερώνεται ο αναγνώστης, ε, ο ενδιαφερόμενος για τη χρηματοδότηση, τι είδους χρηματοδοτήσεις υπάρχουν, τι είδους οργανώσεις χρηματοδοτούνται όλα αυτά τα χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με συνεκτικό τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουμε να συλλέξουμε με σωστό τρόπο τις πληροφορίες. Πολλοί μας είπαν στον τομέα των ΜΚΟ ότι υπάρχουν πολλές πληροφορίες ότι είναι, που είναι διαθέσιμες και δεν είναι ψέμα αυτό, δεν είναι λάθος. Αλλά στην ουσία έχουμε να κάνουμε με ένα πάζλ εδώ διαθεσίμων τμήματων και κομματιών αν κάποιος έχει χρόνο, αν κάποιος έχει ταλέντο, μπορεί να τα συνδυάσει αυτά και να βρει κάποια πράγματα. Ποιος τώρα έχει το χρόνο, ποιος έχει την ικανότητα να το κάνει είναι μια άλλη ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σκεφτήκαμε να ακούσουμε καλύτερα και τις επόμενες τρεις παρεμβάσεις, από χρόνο πάμε καλά, και μετά να γίνουν οι ερωταπαντήσεις. Για να, μην, να, να είμαστε πιο εστιασμένοι. Μπορούμε λοιπόν να ακούσουμε την Επιτροπή το ελεγκτικό συνέδριο και μετά να κάνουμε μία ε, συζήτηση. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο Ζαν Λουιβίλ, διευθυντής στη, Γενική, στη Διεύθυνση Β για την ε, Ανάπτυξη και Μετανάστευση, Γενική Διεύθυνση διεθνισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που διοργάνωσε αυτή τη συζήτηση, πολύ ευπρόσδεκτη. Γνωρίζετε ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν γίνει πολύ σημαντικοί παίκτες και λήπτες κονδυλίων τα τελευταία χρόνια και έχουν νόημα αυτές οι συζητήσεις. Ε, βέβαια, ε, χάνουμε ένα κομμάτι αν εστιάσουμε μόνο στη ΣΜΚΙΟ, Γιατί ε, έχουμε ένα κομμάτι μόνο των χρηματοδοτήσεων στη κοινωνία των πολιτών, το 25%. Γιατί η χρηματοδότηση στη κοινωνία των πολιτών συνολικά είναι πολύ μεγαλύτερη και ανέρχεται σε δύο δις σήμερα μόνο για την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Άκουσα πολύ προσεκτικά και τη μελέτη και τα συμπεράσματα είναι ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τη συζήτηση που κάναμε το 2012 όπου προσπαθήσαμε να πάμε πέρα από τον κύκλο των ΜΚΟ και να δούμε την κοινωνία των πολιτών εν γέννη. Η ΜΚΟ προφανώς και παίζουν μεγάλο ρόλο, αλλά είναι ένα κομμάτι μόνο μιας ευρύτερης εικόνας. Έχουμε επιχειρήσεις, εργοδότες, ε, επιστήμονες, ε, ιδρύματα, ε, συνεταιρισμούς που απαρτίζουν την κοινωνία των πολιτών και παίζουν ενεργό ρόλο στον τομέα της ανάπτυξης. Και αυτό λοιπόν ήθελα να το τονίσω από την αρχή. Άκουσα ότι ένας ενιαίος ορισμός των ΜΚΟ θα βοηθούσε. Το καταλαβαίνω αυτό. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε να το εντάξουμε αυτό στη δουλειά μας και υπάρχει ε, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 15-12 του 12 με βάση την ανακοίνωση της Κομισιόν που εγκρίθηκε και από το Κοινοβούλιο και ο ορισμός αυτός έχει μπει πάλι στον σχετικό κανονισμό που ε, περιλαμβάνει τον ορισμό ως νομικό κείμενο. Ένα άλλο στοιχείο, και μπορώ να σας διαβάσω και τον ορισμό, <clears throat> είναι ευρύς. Δεν είναι νομικός ορισμός καθ' αυτός, γιατί έχουμε διαφορετικές καταστάσεις 28 στα 28 κράτη-μέλη. Αλλά αν δούμε τα στάδια, το νομικό πλαίσιο, το ΜΚΟ, ε, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση γιατί σε κάθε κράτος Υπάρχει ε, ειδική ρύθμιση για τις ΜΚΟ και αυτό μπορεί να δυσκολέψει πολύ κάποιες χώρες όταν γίνεται λόγος για την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθε. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει ε, συλλογική χρηματοδότηση στις ΜΚΟ γιατί χρηματοδοτούμε έργα ε, εστιάζουμε δηλαδή την υποστήριξή μας σε στόχους και αποτελέσματα που σχετίζονται με τις ΜΚΟ και είναι και υπεύθυνε λογοδοτούν οι ΜΚΟ. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένο εταίρο και χρηματοδοτούμε ένα έργο ε, διότι θεωρούμε ε, ότι αξίζει να χρηματοδοτηθεί δεν ε, κρίνουμε τις άλλες δραστηριότητες τους με την προϋπόθεση ότι θα είναι σύνομες και θα ε, ακολουθούν τις διαδικασίες που προβλέπουμε. Και αυτό είναι σημαντικό. Ως παράδειγμα υπάρχουν και άλλα. Ταυτόχρονα ε, ξέρουμε ότι και με το Contract Tandenauer Foundation οι μελέτες δείχνουν ότι θα πρέπει προμήθειες να γίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια, όχι επειδή ανήκουν σε ένα κόμμα ή σε άλλο, αλλά γιατί το ίδιο ισχύει ε, και σε πάρα πολλές άλλες κατηγορίες οργανώσεων. Εάν μία ΜΚΟ λοιπόν έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό, αυτό δεν είναι το κομβικό χαρακτηριστικό κριτήριο που θα χρησιμοποιήσουμε για το αν θα το χρηματοδοτήσουμε ή όχι. Το θέμα είναι αν η δραστηριότητα η οποία ζητείται να χρηματοδοτηθεί, ε, αν θέλετε, συμπίπτει με τους στόχους τους οποίους έχουμε. Οι ΜΚΟ μπορούν να ε, προβάλλουν τα αιτήματά τους, ε, να ζητήσουν υποστήριξη και όχι μόνο. Αν δούμε την ΕΚΟ, την ΤΕΦΚΟ και τι χρηματοδοτούν ως έργα δηλαδή, ε, τα προγράμματα λαμβάνουν χώρα σε πολλές και διάφορες χώρες και επικίνδυνα πολλές φορές περιβάλλοντα. όταν μιλάμε για παροχή ιατρικής βοήθειας ή φαρμακευτικής βοήθειας ή βασικών υπηρεσιών και υποστήριξη σε ανθρώπους στο Χαλέπι ή σε άλλες απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, αυτό μπορεί να το κάνει επιτόπια μία ΜΚΟ, κανένας άλλος. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι αυτά ε, είναι θέματα με τα οποία ευχαρίστως θέλουμε να συνεργαζόμεθα με ΜΚΟ. Τα προβλήματα με τις ΜΚΟ δεν είναι διαφορετικά από ότι όταν συνεργαζόμεθα με άλλες ε, εταιρείε ή ΜΚΟ έχουν χαμηλότερο κόστος όμως από ότι άλλες οργανώσεις. Ό,τι κάνουμε το δημοσιεύουμε, συμβάσεις, ε, δικαιούχους κλπ. Υπάρχει πλήρης διαφάνεια δεν πάμε να ξεφύγουμε από τις υποχρεώσεις μας εις ό,τι αφορά την διαφάνεια ε, στα θέματα αυτά. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας όταν λέτε ότι δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει κατανοητή δράση επιμέρους τμήματων και διευθύνσεων της Κομισιόν, γιατί υπάρχει διαφορετική διοίκηση, αν και οι βασικοί κανόνες είναι οι ίδιοι. Μπορεί να διαφοροποιείται η λειτουργία μας πολλές φορές και υπάρχουν πολλές φορές διαφορές στη λειτουργία. Βέβαια δεν θα αποφασίσω εγώ αν θα έχουμε πιο συγκεντρωτικό σχήμα ε, ή όχι. Αυτό θα αποφασιστεί από τους υπεύθυνους συναδέλφους, υπεύθυνους για αυτό το θέμα. Επίσης αναφέρθηκε ότι υπάρχουν χρήματα που διοχετεύονται σε κονσόρτσια ΜΚΟ και δεν είναι σαφές πού ακριβώς καταλήγουν τα κονδύλια αυτά. Θα ήθελα να θυμίσω κάτι ακόμα, ότι ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει και η Κομισιόν πρέπει να υπογράψει τη σύμβαση με την επικεφαλής ΜΚΟ ενός κονσόρτσιου, αλλά και με τους συμμετέχοντες, δηλαδή Όλα, όλοι οι εταίροι του κονσόρσιου είναι καταχωρημένοι στα συστήματά μας και είναι γνωστοί λοιπόν και κοινοποιούνται τα ονόματά τους υπ' αυτή την έννοια. Καμιά φορά είναι πολύ επαχθές αυτό από διοικητική πλευράς, αλλά όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια, τα κονσόρτσια μπορεί να έχουν 50 ανθρώπους μπορεί, ή 50 οργανώσεις που θα πρέπει να υπογράψουν. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε το σύστημα λειτουργίας. Σταματώ εδώ γιατί ήδη μακρηγόρησα και ευχαρίστως να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βίλ. Ε, ε, ε, βάλατε ένα θέμα ότι γιατί μας απασχολεί αφού είναι όλα αριθμισμένα και κανονισμένα. Εδώ ζητώ την κατανοησή σας στον τομέα αναπτυξιακή βοήθεια ή βοήθεια γειτονίας. Προσπαθούμε να στέλνουμε και αντιπροσωπείες, να κάνουμε επισκέψεις. Υπάρχουν ειδικέ εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, παρακολουθούμε τα θέματα και ενημερωνόμαστε για τα κονδύλια και τους παραλήπτες. Αλλά υπάρχει και μια, ένα νεκρό σημείο, αν θέλετε. Ε, σε αυτό δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και ακριβώς αυτό ψάχνουμε. Και γι' αυτό ζητούμε και τη βοήθειά σας. Γιατί ε, δεν πρέπει να επικριθούμε για το γεγονός ότι θέλουμε ένα πιο κεντρικό, συγκεντρωτικό σύστημα για να παρακολουθούμε την τύχη των κονδυλίων. Το σύστημα θέλουμε να είναι απλό και ένας άνθρωπος με κοινή λογική να μπορεί απ' έξω να δει και να καταλάβει τι γίνεται με τα χρήματα αυτά. Έτσι όπως είναι η οργάνωση αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετείται αυτός ο σκοπός. Γι' αυτό ε, παρακαλώ την κατανόησή σας για το ενδιαφέρον μας, γιατί άλλωστε προασπίζουμε και τα χρήματα των φορολογουμένων μας έτσι. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Στράσερ ε, αναπληρωτής μηματάρχης ε, στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Είχα τη χαρά να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα Live 1420 που είναι για το περιβάλλον και να εξηγήσω γιατί στηρίζουμε και τις ΜΚΟ. Καταρχήν να αναφερθούμε σε, στην ιδεολογική σκέψη 33 του κανονισμού LIFE που αναφέρεται στη Σύμβαση Άρχους για το περιβάλλον και την ε, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Η Σύμβαση υπογραμμίζει το έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και αναφέρεται η ανάγκη για την υποστήριξή τους αφού προβάλλουν και προασπίζονται τις ανησυχίες και τα προβλήματα των πολιτών. Στηρίζεται λοιπόν η εφαρμογή των προγραμμάτων τους, ε, γιατί έτσι υπάρχει και καλύτερη ευαισθητοποίηση για θέματα περιβάλλοντος και κλίματος. Το LIFE Ο κανονισμός LIFE έχει ένα ειδικό άρθρο, το άρθρο 21, που αναφέρεται σε επιχειρησιακή χρηματοδότηση. Στηρίζει δηλαδή ΜΚΟ ε, στο περιβάλλον και το κλίμα, δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και σύμφωνα με το κανονισμό LIFE θα πρέπει να προωθούν και καλύτερη διακυβέρνηση στους δύο τομείς περιβάλλον, κλίμα. Στο πρόγραμμά μας Α, να σας δώσω και κάποια στοιχεία για να δείτε πού βρισκόμαστε. Χρηματοδοτούμε ΜΚΟ με 10 δις ευρώ το χρόνο και συγχρηματοδότηση μπορεί να φτάσει στο 70% στο life. Η Κομισιόν είπε ότι πρέπει να πάει μέχρι το 60% το ποσοστό της συγχρηματοδότησης. Πώς επιλέγουμε τους εταίρους της ΜΚΟ. Κάθε δύο χρόνια γίνεται ε, μια δημοσίευση ε, πρόσκλησης ε, για εκδήλωση ενδιαφέροντος τον Απρίλιο του 2017 θα γίνει για τα τελευταία για τα επόμενα δύο χρόνια. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος και προτάσεων γίνεται δημόσια, η επιλογή επίσης με μεγάλη διαφάνεια. Έχουμε κριτήρια επιλεξιμότητας, συμβασιοποίησης, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες, θα πρέπει να ε, ε, επιδιώκουν το κέρδος, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον και το κλίμα και να έχουν, να ε, έχουν ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή να συνεργάζονται με τρεις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ε, ΜΚΟ. Έχουμε και εμπειρογνώμονες εξωτερικούς για να μας βοηθούν στη διαδικασία επιλογής η οποία μετά γίνεται στην αρμόδια επιτροπή. Τώρα για τις ΜΚΟ ε, έχουμε ε, περίπου 66 ε, είχαμε προτάσεις και επιλέξαμε 32 ΜΚΟ. Σε από πού επελέγησαν 65% στην περιβαλλοντική πολιτική και οι υπόλοιποι στην, από το τομέα του κλίματος. 38% εργάζονται στην βιοπικιλότητα, 28% ε, στο κλίμα, τα θέματα δηλαδή που καλύπτονται από τις 32, 9% είδωρ, γεωργία 9%, απορρίμματα, απόβλητα 6%. Τέλος θα ήθελα να αναφέρω και την ιστοσελίδα μας του Life που είναι πολύ εύκολο να την βρείτε. Ε, εκεί υπάρχει μία σύνοψη των επελεγμένων έργων live ε, με μεγάλη διαφάνεια. Εδώ και 15 χρόνια οι όπου που ε, είχαν επιλεγεί υπάρχουν και μπορείτε να τις βρείτε. Ε, υπάρχει ε, ευρύτερη υποστήριξη από το LIFE. Γιατί? Γιατί η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη και νομικά να υποστηρίζει τις ΜΚΟ αφού αυτό προβλέπεται και στον κανονισμό LIFE. Δεύτερον, η Κομισιόν χαιρετίζει αυτή την υποχρέωση, ε, δηλαδή να προωθήσει καλύτερη διακυβέρνηση στο περιβάλλον και το κλίμα μέσα από την υποστήριξη αυτών των ΜΚΟ που επιλέγονται με δίκαιο τρόπο και με τρόπο διαφανή. Η επιλογή θέλει να ενισχύσει την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε μια διαδικασία μέσα από διάλογο σε θέματα ε, περιβάλλοντος και κλίματος περιμένουμε από τις ΜΚΟ να υποστηρίξουν ε, τη δράση τους ε, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση ε, και να ε, παίξουν το ρόλο του θεματοφύλακα στον τομέα της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της συμμόρφωσης και βεβαίως συμβάλλουν και επιστημονικά μέσα από ε, επιστημονικές μελέτες και πραγματογνωμοσύνη. Αν μου επιτρέπετε θα επανέλθω σε κάποια κριτική που ακούγεται ξανά και ξανά στα πλαίσια της χρηματοδότησης των ΜΚΟ. Μία κριτική που ακούμε είναι η εξάρτηση ότι οι ΜΚΟ δηλαδή παίρνουν χρηματοδότηση και δεν έχει υποχρέωση σε σχέση με επιχειρησιακή ανεξαρτησία. Όχι. Ε, η ΜΚΟ που υποστηρίζονται στα πλαίσια του LIFE έχουν και τη δυνατότητα να εκφράζουν την, τις απόψεις τους στα πλαίσια της πολιτικής μας. Ε, υπάρχει ε, χρηματοδότηση για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία τους, είναι ελεύθερες να εκφράζουν απόψεις και τις εκφράζουν ως ε, διαδικασία του δημοκρατικού διαλόγου. Εμείς στηρίζουμε τις ΜΚΟ ε, για να εκφράζονται ελεύθερα. Αυτό είναι η πεμπτουσία της πολιτικής μας ε, απέναντι στη ΜΚΟ. Καμιά φορά ακούμε ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας. Εγώ σας παραπέμπω στην ιστοσελίδα του Live που αναφέρονται οι προκηρύξεις, τα κριτήρια ευδιάκριτα, ξεκάθαρα και αναφέρονται και οι επιβελεγμένες ε, ΜΚΟ. Όλες αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η διαδικασία επιλογής των ΜΚΟ ε, γίνεται με τρόπο διαφανή. Σε άλλους τομείς ε, ακούγεται η κριτική ότι υπάρχει έλλειψη ελέγχου. Εμείς στο live επιλέγουμε τις ΜΚΟ με βάση τη σημασία που έχουν για τις πολιτικές μας, τη δυναμική που έχουν να επηρεάσουν ε, την ευρωπαϊκή πολιτική και τα μέσα που διαθέτουν για την εφαρμογή. Η ΜΚΟ ε, ανταποκρίνονται σε ένα πρόγραμμα εργασίας συμφωνημένο το οποίο παρακολουθείται και επαληθεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παληθεύομαι ότι τηρούνται οι κανόνες που έχουν τεθεί στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κομισιόν δέχεται τις ε, διαφορετικές απόψεις. Οι απόψεις οι διαφορετικές επηρεάζουν θετικά την πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα. Ε, εν προκειμένου στα πλαίσια του προγράμματος LIFE. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στράσερ. Είναι πολύ ενδιαφέρον που μιλήσατε για ε, λειτουργικές δαπάνες, ε, στόχοθετημένες δράσεις ε, που συμφωνούνται. Δεν ξέρω ε, πώς γίνονται αυτές οι συμφωνίες και αν υπάρχουν αντιθέσεις μέσα στους κόλπους της Κομισιόν. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει συμφωνία για συγκεκριμένους στόχους που μπορεί να ε, ακολουθούν συγκεκριμένες ενδεχομένως και κομματικές πολιτικές. Δηλαδή σε ποιο βαθμό ε, ισχύουν αυτές οι συμφωνίες. Μπορεί δηλαδή να ε, ανοίγεται πεδίο για τους λόμπιστς εδώ. Ε, πάντως ε, σας ευχαριστώ πολύ για την συμβολή σας που νομίζω ότι εξυπηρετεί την καλύτερη διαφάνεια. Πάμε τώρα στο ελεγκτικό συνέδριο. Ο κύριος Ντένις Βέρνερους ε, ασχολείται με τη ΣΜΚΙΟ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Το ελεγκτικό συνέδριο σας ευχαριστεί για την πρόσκληση. Τονίζω και εγώ πριν αρχίσω στα αγγλικά την παρουσίασή μου ότι η παρουσίαση αυτή ασχολείται με την παγκόσμια Ευρώπη, Global Europe, και δεν αναφέρεται στις ΜΚΟ στα κράτη-μέλη που δραστηριοποιούνται εκεί και χρηματοδοτούνται ενδεχομένω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κυρίως ελέγχει ε, της ε, επιλεγής σε μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, όσον αφορά τους νόμιμους ε, οικονομικούς ελέγχους και το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων βρίσκονται υπό το κεφάλαιο Global Europe της ετήσιας έκθεσής μας. Επίσης ε, και στις ετήσιες ε, εκθέσεις CDF e και σε κάποιες ειδικέ εκθέσεις τις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ ε, σήμερα. Πρόκειται για τις εκθέσεις επιδόσεων τις οποίες κάνουμε σε σχέση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το 2009 είχαμε ε, την αξιολόγηση της ε, ε, διαχείρισης της Κομισιόν των Non-State Agents Επίσης, ε, λίγο αργότερα, πάντα το 2009, ε, δημοσιοποίησαμε μία έκθεση σχετικά ε, με την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών. Είχαμε την έκθεση του 2012 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ε, τροφική ασφάλεια ε, στην υποσαχάρια Αφρική. Κυρίως δε αναφερθήκαμε στη δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων κατά την έννοια αυτή και πιο πρόσφατα το 2015 είχαμε και την, τον έλεγχο EIDHR σχετικά με την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωσης ε, για την ε, ε, καταπολέμηση των βασανισμών και την κατάργηση της θανατικής ποινής. Στα πλαίσια της εργασίας μας αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ορίσουμε ε, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις πριν ξεκινήσουμε δηλαδή τον ε, οικονομικό τους ε, έλεγχο. Πολλά έχουν γραφτεί και υποθεί σχετικά με τον ορισμό, ακόμα και σήμερα έγινε μια σχετική αναφορά. Ε, ε, μιλάμε για οργανώσεις που δεν είναι ε, Ηνωμένα Έθνη, που δεν είναι εθνικές οργανώσεις, αυτές δεν ορίζονται ως μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αναφερόμαστε σε μη κρατικές οργανώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται ως, αναφέρονται ως NGO ή CSO. Έχουμε επίσης ε, και την ε, απόφαση, μια σχετική απόφαση η οποία ε, ορίζει τι δεν είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Η χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων ενέχει κάποιους ε, κινδύνους. Βεβαίως ε, από ε, οικονομική άποψη και από άποψη οικονομικής διαχείρισης πάντα υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Ορισμένοι από αυτούς τους κινδύνους συνδέονται και σε πολλές περιπτώσεις και σε οργανώσεις οι οποίες δεν ορίζονται ως διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι τοπικές. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν αντιμετωπίζονται προβλήματα σε αναπτυσσόμενες χώρες ε, όπου εμπλέκονται μη, τοπικές μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις. Επίσης ε, έχουμε πολλέ συναλλαγέ και γενικές ή σχετικές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μέσω πολύ περίπλοκων αλυσίδων ας πούμε οργανισμοί Ηνωμένων Εθνών οι οποίε υλοποιούν τα προγράμματά οι οποίοι υλοποιούν τα προγράμματά του μέσω ε, μη κυβερνητικών ε, ε, οργανώσεων. Έχουμε επίσης και 8 διαφορετικά εργαλεία συνεργασίας από το 2014 μέχρι το 2020 και σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση. Ε, όπως ε, ακούστηκε και προηγουμένως, ε, η χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, μπορεί να γίνει μέσα από grants ή μέσα από συγκεκριμένες συμβάσεις, service contracts ε, σε κάθε περίπτωση πάντως το θέμα ε, ε, της, του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι αυτό το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται η υπόψη. Η Κομισιόν γνωρίζει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και γνωρίζει ότι κυρίως βασίζονται στις δικές τους δηλώσεις self-declaration καθώς επίσης και στη μεθοδολογία ελέγχου που έχουν οι γενικέ διευθύνσει ε, της ε, Κομισιόν. Ε, Επίση, υπάρχουν και τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στο κοινό σύστημα πληροφόρηση RELEX, στο CRIS. Γνωρίζουμε βέβαια ότι οι πληροφορίε αυτές δεν είναι πλήρε και επομένως θα πρέπει να βελτιωθούν περισσότερο. Ε, όσον αφορά τώρα τους κινδύνους ε, νομιμότητος, ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά, τους, όσον αφορά τα grants, όσον αφορά αυτά τα, τα δάνεια. Κυρίως ο κίνδυνος σχετίζεται με μη επιλέξιμες δαπάνες ε, αυτή τη στιγμή ε, βεβαίως το πρόβλημα εντοπίστηκε γενικά ε, στο, στο γενικό πλαίσιο των ελέγχων που κάνουμε για τις αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές δαπάνες οι οποίες δεν έχουν άμεση σχέση απαραίτητα με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Έλεγα λοιπόν ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα, πολλές φορές τα έντυπα δεν είναι σωστά, πολλές, σε πολλές φορές λείπουν κάποια στοιχεία όταν έχουμε ε, συμβάσεις σε πολλές ε, περιπτώσεις ε, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με, τις, με τους εξειδικευμένους όρους του συμβολέου. Ε, ε, για τις ε, περιπτώσεις ελέγχου συμμόρφωσης βεβαίως θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε ακόμα περισσότερο επί της ουσίας να δούμε δηλαδή εάν κάποια μη κυβερνητική οργάνωση δεν εκπροσωπεί στην ουσία κάποια ιδιωτικά συμφέροντα ή κάποια κυβερνητικά συμφέροντα. Τώρα έχουμε το θέμα της ε, ορατότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι ένα προβληματικό στοιχείο. Δεν είναι τόσο ε, συγκλονιστικό, αλλά να μην λησμονούμε ότι πρόκειται για ε, δάνεια και να μην λησμονούμε επίσης ότι πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις ζουν και δρούν χάρη στην ενωσιακή χρηματοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να είναι πιο ορατή αυτή η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές δεν βλέπουμε καν καν ε, τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αναφορά στην συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, έχουμε διαπιστώσει επίσης και κάποιους κινδύνους όσον αφορά τις επιδόσεις. Ας πούμε σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εμπλοκές με κυβερνητικές οργανώσεις. Κυρίως διαπιστώσαμε τέτοια προβλήματα στα προγράμματα για την τροφιμική ασφάλεια στην υποσαχάρια Αφρική. Επίσης, ε, όταν είναι πολύ μικρή η χρηματοδότηση και κατακαιρματίζεται σε πολλά μικρά, ε, προβλή, σε πολλά μικρά projects, ε, τότε έχουμε αυτό το, αυτόν τον κατακαιρματισμό που δημιουργεί προβλήματα, γιατί στην ουσία από τη στιγμή που μιλάμε για πολλά μικρά προγράμματα και πολλές μικρές χρηματοδοτήσεις, η απόδοση είναι πάρα πολύ μικρή. Ε, στους κινδύνους ε, που σχετίζονται με τις ε, επιδόσεις διαπιστώνουμε και προβλήματα όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων. Δηλαδή η Κομισιόν δεν γνωρίζει πάντα τον τον δικαιούχο ε, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κυρίως όταν ενέχονται πολλές μικρές και τοπικές ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν ε, την, την ικανότητα που έχουν οι πιο μεγάλες οργανώσεις. αυτό το αναφέραμε και στην έκθεσή μας του 2009. Ε, και επίσης ε, έχουμε και τα άμεσα κόστη τα οποία μπορεί να αποτελούν και το 7% ε, βάσει του άρθρου 124 παράγραφος 4. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, ειλικρινά πρέπει να πω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί για τα διαρθρωτικά ταμεία πολύ σωστά προβλέπεται shared management, κομισιόν κράτη-μέλη, ενώ σε προγράμματα που γίνονται ε, ε, με τις ΜΚΟ, εκεί δεν δραστηριοποιείστε. Γιατί αυτό είπατε στην αρχή. Δεν το χωράει το κεφάλι μου δηλαδή αυτό. Ε, είναι ένα μεγάλο κενό, όπου το ελεγκτικό συνέδριο θεωρώ ότι θα έπρεπε να αναλάβει ευθύνη. Μπορεί να αποτελέσει αυτό ένα σημείο στην έκθεσή μου, ώστε να απαντηθούν κάποια ερωτήματα. Λοιπόν, καλώς. Ε, θα κάνουμε τώρα τη συζήτηση. Όλοι όσοι είναι εδώ μπορούν να κάνουν ερωτήσεις στην Κομισιόν, στο ελεγκτικό συνέδριο ή στους εμπειρογνώμονες. Έχω ήδη δύο εγγεγραμμένους ομιλητές, αλλά θα ήθελα να σας καθησυχάσω διότι αμέσως θα δώσουμε το λόγο στη ΜΚΟ και μετά θα ακολουθήσει πάλι μισάωρη συζήτηση. Οπότε τώρα κάντε ερωτήσεις προς την Κομισιόν, τους εμπειρογνώμονες και το ελεγκτικό συνέδριο. Ο κύριος Ντες, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι από την αρχή παρόν, αλλά ακούσαμε ενδιαφέρον ό,τι ακούσα. Έχω ερώτηση στην Κομισιόν και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Γιατί αντιμετωπίζω τόσο διαφορετικά τα ε, ευρωπαϊκά κονδύλια. Εγώ είμαι, ε, δραστηριοποιούμε στην αγροτική πολιτική και Ξέρω περιπτώσεις ε, όπου επευλήθησαν πρόστιμα ε, διότι δεν υπήρχε μεγάλη διαφάνεια στην λειτουργία των ε, εκμεταλλεύσεων, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. γιατί δεν ισχύει αυτό σε όλους τους τομείς. Υπάρχει έλλειμμα εδώ. Ένας γεωργός όταν παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λογοδοτεί 100%. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις ΜΚΙΟ. Πρέπει να ε, υπάρχει στο διαδίκτυο ποιος πήρε πόσα χρήματα με αυστηρότητα όπως τη Γεωργία. Τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, παρακολουθούνται και να ε, υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και για τις ΜΚΟ. Είναι πολύ σημαντικό. Το έχω πει και στο Στρασβούργο. Πολλέ φορέ έχω ρωτήσει ποιος τις χρηματοδοτεί. Πώς νομιμοποιούνται να δραστηριοποιούνται. Ποια είναι, ποιος είναι ο κατάλογο των μελών τους. ποιο είναι ο ισολογισμό τους, ε, έσοδα, δαπάνες. Ε, όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν αλλιώ. Δεν μπορεί να υπάρχει διαφάνεια. Δεν μπορεί να νομιμοποιείται η δράση τους. Βεβαίω, ε, δεν, ε, μην με παρεξηγήσετε, υπάρχουν και πολύ καλέ ΜΚΟ, αλλά δεν θέλω να χρηματοδοτούνται ΜΚΟ από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που ακολουθούν μη, συμφωνημένου στα πλαίσια της πολιτικής μας ε, στόχους. Δεν μπορούμε να δαπανούμε τα χρήματα των φορολογουμένων για αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ. Αυτή είναι ερώτηση που θα απαντήσει και το ελεγκτικό συνέδριο και ο κύριος Στράσερ ενδεχομένως. Αλλά όχι ακόμα, παρακαλώ, ας ακούσουμε και τις επόμενες ερωτήσεις. Ε, ο κύριος Γιάβορ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίαση της Επιτροπής. Ευχαριστώ και αυτούς που συνέταξαν τη μελέτη και το ελεγκτικό συνέδριο. Θα προσπαθήσω να είμαι ψύχρεμος σε αυτή τη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση περίπλοκη. Έρχομαι από μια χώρα όπου οι ΜΚΟ πιέζονται συνεχώς από την ίδια τη κυβέρνηση με διαφορετικούς τρόπους, διοικητικούς, ποινικού, εκστρατείες παραπληροφόρησης κτλ. Βρίσκομαι λοιπόν σε κάπως ευαίσθητη κατάσταση όταν μιλάω για τις ΜΚΟ ξεκινώντας να πω ότι στα πλαίσια της μελέτης που έχουμε μπροστά μας ε, τη νιώθω λίγο ατελή και σχετικά προκατελημένη. Γιατί το λέω. Εγώ είμαι υπέρ ε, της πλήρους διαφάνειας σε όλους τους τομείς και για τις ΜΚΟ και για τις μεγάλες επιχειρήσεις και για τη δημόσια διοίκηση. Να είμαι ειλικρινής. Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της μελέτης δεν μου δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Είναι λογικές οι προτάσεις αυτές και νομίζω ότι και σχετικά εφαρμόσιμες. Ένας καλύτερος ορισμός των ΜΚΟ, γιατί όχι. Οι ΜΚΟ το θέλουν αυτό και αν δεν είναι ικανοποιημένες μπορούν να το κάνουν, να το δείξουν αυτό μέσα από τις κυβερνήσεις τους. Νομίζω επίσης ότι και μια καλύτερη δημοσιοποίηση και δημοσίευση των στοιχείων για τις ΜΚΟ είναι θετικό. Τα περισσότερα από τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε επίπεδο κράτους μέλους και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα δεν είναι λοιπόν η έλλειψη των στοιχείων των δεδομένων από τις μικιό, αλλά ο τρόπος που τα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δημόσιες διοικήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη συμμοσίευση αυτών των δεδομένων. Είμαι υπέρ επίσης και της, ε, του ελέγχου και της ανάληψης ευθύνης. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημά μας εδώ δεν είναι η ΜΚΟ βέβαια, τα χρήματα που δίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνούν ίσα ίσα το ένα δις. Αν δει κανείς τι κάνουμε στην κοινή αγροτική πολιτική, στην οποία αναφέρθηκε ο Ντες, δεν υπάρχει σχέση. Το θέμα λοιπόν δεν είναι το ύψος του ποσού. Δεύτερον, τα χρήματα τα οποία δαπανά κάθε ΜΚΟ ελέγχονται και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Υπάρχουν απαιτήσει από τις κοινέ διαχειριστικές αρχές, από τις εξωτερικές υπηρεσίες της Επιτροπής. Εγώ συνεργάζομαι με ΜΚΟ και βλέπω το γραφειοκρατικό βάρος το οποίο πρέπει να εξυπηρετήσουν. Ίσως για το κοινό αυτή η προσπάθεια να μην είναι απολύτως διαφανής, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Έχω κάποια θέματα επίσης και με τους βασικούς στόχους της μελέτης. Ο τίτλος λέγει «Δημοκρατικός έλεγχος και δημοσιονομικός έλεγχος των ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό». Ε, μετά στην τελευταία σελίδα λέγεται η διαμόρφωση των πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι ποιος ελέγχει ποιον εδώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ποιος επηρεάζει κυρίως τη λήψη των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν παράδειγμα. Δεν ξέρω αν ο Επίτροπος Έτιγκερ σαν παράδειγμα στο λόμπι το οποίο τον περιβάλλει παίρνει πληροφορίες και συναντάται περισσότερο με την Deutsche Telekom παρά με όλες τις ΜΚΟ. Οι συναντήσεις που έκανε με την Deutsche Telekom είναι περισσότερες. Συνεπώς λοιπόν το ποιος επηρεάζει τις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτείτε. Υπάρχουν και κάποιες ελάσσονες παρατηρήσεις αλλά δεν έχω άλλο χρόνο πια. Ίσως ένα πράγμα μόνο για την χρηματοδότηση των ΜΚΟ και οι δύο από τις πέντε μελέτες αφορούν σε ΜΚΟ που δεν χρηματοδοτούνται περίεργως από την Ένωση. Οπότε διαρωτώ με λιγάκι εδώ ε, ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της έρευνας. Και μια τελευταία ερώτηση. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να βρούμε προβλήματα με τις ΜΚΟ, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει πρόβλημα με την χρηματοδότηση, η δυσκολία πρόσβαση στη χρηματοδότηση, οι μικρές ΜΚΟ που δεν μπορούν να πάρουν χρήματα λόγω ακριβώς των υψηλών επιπέδων ελέγχου και γραφειοκρατίας που δημιουργεί προβλήματα για τις ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ που είναι συστατικό της δημοκρατίας βασικό δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Επίσης υπάρχουν μεγάλες χρηματοδοτικές προσπάθειες τις οποίες δεν μπορούν να ωφελήσουν τις μικρές μικιό. Και τέλος, κάτι που λείπει είναι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που οργανώνονται από τις ίδιες τις κυβερνήσεις. Νομίζω ότι αυτές είναι κάτι το αντίθετο με την κοινωνία των πολιτών και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν τέτοιες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλά μένει να γίνουν λοιπόν εδώ, αλλά δυστυχώς δεν είναι και τόσο αυτά που περιλαμβάνει η έρευνα. Ε, αγαπητοί μου, βλέπω ότι φέρατε και φαν μαζί σας ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο ομιλητή, δεν θα βγάλω λόγο, αλλά θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στα θέματά μας. Είναι λυπηρό για το φορολογούμενο ε, το σύστημα που υπάρχει. Καταρχήν, που είναι ο ορισμός της ΜΚΟ. Είναι πολύ διάτρητος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις διάφορες γενικές διευθύνσεις βλέπουμε πόσο διαφορετικά γίνονται τα πράγματα, ε, δηλαδή οι νομικοί κανόνες διαφέρουν. Και όταν ε, πρόκειται για διάθεση κονδυλίων σε τρίτους, τότε οι εμπειρογνώμονες μιλάνε για μαύρο κουτί. Η τερα δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν τα λεφτά και δεν είναι αυτό σωστό μήνυμα για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για απλό, απλούστευση. Μια χαρά, ποιος θα διαφωνούσε. Θέλουμε και ηλεκτρονικές ε, ε, προτάσεις, ψηφιοποίηση και οι διατάξεις θα πρέπει να εναρμονιστούν. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι πρέπει να γίνουν ενιαίες οι διατάξεις, αλλά θα πρέπει να ε, εφαρμόζεται με νέο τρόπο το δίκαιο, οι νομικοί κανόνες. Και τι κάνει η Κομισιόν ε, γι' αυτό, όχι μόνο για την εναρμόνιση των διατάξεων, αλλά μεταξύ των γενικών διευθύνσεων να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο, γιατί μόνο τότε έχουμε ενιαίο νομικό καθεστώς. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ ένας κυρίος από το κοινό μας που είχε δηλώσει το... ότι ήθελε να λάβει το λόγο από την αρχή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Καρλ Ντόνιν και είμαι διευθυντής της Διεθνούς Διαφάνειας στο Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφάνεια, η λογοδοσία είναι πολύ σημαντική για μας προκειμένου περί δαπανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να δούμε τις δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων και την ε, διαφάνεια και τη λογοδοσία εκεί. Αυτά τα θέματα είναι οριζόντια, ε, αφορούν όλες τις δαπάνες. Ένα παράδειγμα που αναφέρεται και στην έκθεση, θα πω, που αναφέρθηκε και από τον Πρόεδρο, δηλαδή από τα κονσόρτσια, πώς περνούν τα κονδύλια και από τους εταίρους των κονσόρτσια και φάνουν στις μικρές ΜΚΟ. Ε, έχουν, υπάρχουν κονσόρσια στα πανεπιστήμια στο ε, πρόγραμμα 2020, ε, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο, μέσα από το Ταμείο Ανάπτυξης. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν αυτούς που έκαναν τη μελέτη, σε ποιο βαθμό είδατε ότι αυτά τα θέματα είναι σημαντικά, δηλαδή μπορεί, είδατε διαφοροποίηση Μπορεί η ΜΚΟ καμιά φορά να λειτουργούν καλύτερα από ότι τα πανεπιστήμια, οι ΜΜΕ, οι δημοσίες αρχές, οι εταιρείε συμβούλων ή οποιοδήποτε άλλοι παραλήπτες κοινωτικών ευρω... Ε, ενωσιακών κονδυλίων. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πρέπει δυστυχώς να κλείσουμε το κατάλογο των ε, ομιλητών. Μετά θα ακολουθήσει κι άλλος γύρος ερωτήσεων. Ε, η συνάδελφος Πιτέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, που μου δώσατε το λόγο, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ακούμε και ξανακούμε ότι δεν υπάρχει ορισμός ε, για τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, και ότι αυτό ισχύει, συμβαίνει γιατί είναι, πολλές και είναι πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί στα κράτη-μέλη. Πρέπει να σας πω ότι στην Πολωνία εγώ ήμουν επικεφαλής μιας μη κυβερνητική οργάνωσης και επομένως θα ήθελα να καταλάβω ε, τι εννοείται ας πούμε ε, να μην έχουν και κερδοσκοπικό σκοπό γιατί στην Πολωνία έχουμε δύο ειδών ε, μη κυβερνητικέ ε, ε, οργανώσει. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες έχουν και οικονομική δραστηριότητα. Ρωτώ λοιπόν πώς μπορούμε να ορίσουμε ότι κάποια οργάνωση η οποία ζητά την χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα γιατί γιατί ε, διατρέχουμε τον κίνδυνο να δίνουμε χρήματα τα οποία δεν θα ελέγχουμε που δίνονται και με ποιο τρόπο θα πανώνται. Επίσης, ε, υπό τον γενικό όρο μη κυβερνητική οργάνωση ε, ενδεχομένως μπορεί να κρύβεται μια ομάδα ε, λόμπι. Αυτό έχει συμβεί και στην Πολωνία όπου κάποιες οργανώσεις θεωρούνται μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά στην ουσία, στην ουσία έκαναν δραστηριότητα λόμπι υποβοηθούμενοι και από μέλη του Κοινοβουλίου. Θέλω λοιπόν να μάθω λεπτομερώς πώς πώς προστατεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, απέναντι σε καταχρήσεις και απάτες. Ευχαριστώ. Και αυτή είναι ερώτηση για την Κομισιόν. Λοιπόν, ο... θα απαντήσουν αργότερα οι συνάδελφοι. Ο κύριος Τέρεκ Φόρμεντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς άκουσα πολύ λίγο τμήμα των ε, παρουσιάσεων. Πάντως πρέπει να σας πω ότι το 2009 γνωρίζω την κατάσταση γιατί ήδη το 2009 εγώ ήμουν υπεύθυνος για τον έλεγχο των συμβάσεων με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στην ε, Ουγαλία ε, και τους ε, βοηθούσα εξ της Κομιτείας ε, στην διεκπαιρέωση των προγραμμάτων και λοιπά Δηλαδή κάναμε παροχή υπηρεσιών βάσει των προγραμμάτων και μιλάμε για προγράμματα για βοήθεια παιδιών και για τέτοιου είδους κοινωνικά ζητήματα. Μερικές φορές, και αυτό με εντυπωσίασε, μερικές φορές φορές δεν υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου του τρόπου με τον οποίο είχαν ταπανηθεί τα χρήματα από την μη κυβερνητική οργάνωση. Ε, δηλαδή, ε, Ε, ήταν μάλλον εύκολο να δει κανείς πού έχουν δαπανηθεί τα χρήματα, αλλά πολύ δύσκολο το να ορίσει κανείς την αποτελεσματικότητα της χρήσης των κονδυλίων αυτών. Το ίδιο ε, συμβαίνει και με την ε, ενωσιακή χρηματοδότηση. Δηλαδή, ναι, η μέτρηση των αποτελεσμάτων είναι κάτι δύσκολο. Είπατε και εσείς ότι θα πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις Κομισιόν και στο ελεγκτικό συνέδριο συνέδριο. Ρωτώ λοιπόν να μιλάμε διαρκώς και όλο και περισσότερο για την αποτελεσματικότητα και την μέτρηση της αποτελεσματικότητας. Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις στο μέλλον έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι καλά χρησιμοποιούνται τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα και με τις ίδιες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δηλαδή οι ίδιες να μας πούν πώς είναι δυνατόν να αποδείξουν όχι ότι απλά χρησιμοποιούν σωστά ε, με, με νόμιμο τρόπο δηλαδή τα, τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ε, ότι είναι αποτελεσματική η χρήση αυτή. Ο Σιάνφος Τζέλλερ. Τελευταίος ο μιλητής. Ευχαριστώ. Μια ΜΚΟ είναι μια οργάνωση θεωρώ που εκτός κρατικών δομών και κυβέρνησης αναλαμβάνει δράση και αυτό γιατί δεν θέλει να εξαρτάται από την κυβέρνηση. Σε μία επίσκεψη στις ΕΙΠΑ διαπίστωσα ότι οργανώσεις που ε, ορίζονται ως ΜΚΟ ε, δραστηριοποιούνται για να βοηθήσουν τους αστέρους να βοηθήσουν τους ε, ε, ενοικιαστές. Θέματα δηλαδή που σε εμά τα αναλαμβάνει το κράτος, τουλάχιστον έτσι είναι στη Γερμανία το σύστημα. Και όταν ρώτησα τι επιχορηγήσει παίρνετε από το δημόσιο προϋπολογισμό για να τα κάνετε όλα αυτά, ε, με κοίταξαν κατάπληκτοι και μου είπαν Πώς το σκεφτήκατε ότι ε, παίρνουμε λεφτά από το κράτος. Εμείς προσφέρουμε υπηρεσίες στον κόσμο γιατί δεν ανταποκρίνεται το κράτος στα, ε, στις υποχρεώσεις του. Δεν έχει. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν, δεν μπορεί να τα κάνει το κράτος και εκεί παρεμβαίνουν οι οργανώσεις αυτές. Και ε, μπορούν και να χρηματοδοτούνται εδώ σε εμάς. Όταν όμως ε, υπάρχουν όμως Μικιό που λένε ότι είναι Μικιο και που χρηματοδοτούνται με κρατικά κονδυλία για να παρεμβαίνουν σε πολιτικές διαδικασίες. Α, εδώ ε, υπερβαίνουν τα όρια. Ή θα είναι Μικιο ή θα είναι ε, εταιρεία που διαχειρίζεται πολιτικά συμφέροντα. Εκεί πολλές φορές ε, η ε, οριοθέτηση δεν είναι σαφής και πρέπει να τα διαχωρίσουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ. ακούσαμε πολλές ερωτήσεις. Προτείνω να... Βέβαια θα απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες, το ελεγκτικό συνέδριο, ο κ. Στράσερ για την Κομισιόν και ο κύριος Πανικάλη. Ποιος άλλος ζητεί το λόγο από τους ομιλητές. Γιατί αλλιώς θα απαντήσουν αυτοί που ανέφερα. Πρώτα το ελεγκτικό συνέδριο. Η χρηματοδότηση των ΜΚΟ στον τομέα της αναπτυξιακής ανθρωπιστικής βοήθειας γίνεται κυρίως μέσω άμεσης διαχείρισης. Για το ελεγκτικό συνέδριο αυτού του είδους η δημοσιονομική λειτουργία παρουσιάζει λιγότερους κινδύνους από ότι στα τα ταμεία ή στα ταμεία τη Γεωργία. Οι έλεγχοι είναι εντατικοί, γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τα κεντρικά της Επιτροπής, από τις αντιπροσωπείες σε διάφορες χώρες και τέλος υπάρχει άμεσος έλεγχος ε, της δαπάνης. Τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει και το είπα αυτό είναι η πρόσβαση στα δεδομένα, οι διαφορές συστημάτων ανάμεσα στις γενικές διευθύνσεις και οι δυσκολίες που δημιουργούνται λόγω του ετερογενούς τοπίου που έχει σχεδιαστεί, οκτώ διαφορετικά ταμεία. Η τοπική γεωγραφία λειτουργίας είναι καθοριστική. Αυτά τα εμπόδια λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση του κινδύνου. Έχουμε ακριβώς γι' αυτό το λόγο και εκτός της συγκεκριμένης εκθέσεως για το 2009 δημοσιεύσει ένα έλεγχο λογιστικό επιδόσεων ειδικό για τις ΣΜΚΙΟ γιατί όπως είπα ο κίνδυνος ο οποίος έχει διαπιστωθεί από την παλιά μας εμπειρία είναι υψηλός για τις ΜΚΟ, αλλά όχι μόνο και για άλλους δικαιούχους ποσών. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι το συνολικό ποσό για το MFF Global Europe που πηγαίνει στις ΜΚΟ είναι ένα μικρό τμήμα, ε, πραγματικά πολύ μικρό του κοινοτικού προϋπολογισμού. Νομίζω λοιπόν τα πράγματα εδώ να ξεκαθαρίζονται λίγο και εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να ξεκινήσουμε εμείς ελέγχους επιδόσεων σε συγκεκριμένους τομείς, φυσικά να το κάνουμε. Και ακριβώς οι πρόσφατες εκθέσεις μας λαμβάνουν υπόψη τέτοιου είδους επιθυμίες. Ευχαριστώ. Προτείνω τώρα να απαντήσει ο κ. Στράσερ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Αναφέρομαι σε κάποιες ερωτήσεις που ακούσαμε εδώ. Με ποιους εργαζόμεθα στο πρόγραμμα LIFE, με ποιες ΜΚΟ. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι πολύ αυστηρά. Θέλουμε ε, έκθεση ετήσια για τις δραστηριότητες της ΜΚΟ, να ξέρουμε τι έχει κάνει. Επίσης θέλουμε ισολογισμούς, να ξέρουμε τα οικονομικά τους, είναι ανεξάρτητες, είναι μη κερδοσκοπικές όντως, επίσης ε, η δομή των μελών, με λεπτομέρειες, ποια είναι τα μέλη της οργάνωσης. Και στη φάση της προκήρυξης ζητούμε τις προτάσεις των ΜΚΟ στα πλαίσια ενός προγράμματος εργασίας, το οποίο επίσης είναι ε, κοινό, είναι δημόσιο, δημοσιεύεται. Ε, ε, θέλουμε από εκεί να δούμε ότι εστιάζουν στο περιβάλλον και το κλίμα. Επίσης, ε, πρέπει να δούμε την ανεξαρτησία ή εξάρτηση. Ε, η συγχρηματοδότηση είναι 60% maximum, αλλά από τις 32 ΜΚΟ είναι κάτω από το, 30%, από το 60%. Έχουμε συγχρηματοδότηση ορισμένης 25% και στα κριτήρια επίσης. Εξετάζουμε πολύ προσεκτικά η ΜΚΟ να δραστηριοποιούνται και σε εράνους, ε, ε, ε, δηλαδή για συλλογή κονδυλίων. Να μην εξαρτώνται μόνο από τα, από τα ενωσιακά κονδύλια, αλλά να μπορούν να συγκεντρώνουν και άλλα κονδύλια από άλλες πηγές. Αυτό είναι σημαντικό για την διατηρησιμότητα της δράσης τους. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Ευχαριστώ κύριε Στράσερ για τις διευκρινήσεις από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ, ο κύριος Πανιγκάλη. Ευχαριστώ. Είμαι ο Μάρκο Πανιγκάλη, τμήματάρχη στη DG ΕΚΟ υπεύθυνος για προϋπολογισμό, χρηματοδότηση και έλεγχο. Νιώθω ότι υποχρεώνομαι, αν θέλετε, να σταθώ σε κάποια από τα θέματα τα οποία έθεσαν οι ομιλητές. Κάποιες απαντήσεις δόθηκαν ίσως από άλλους ομιλητές εν μεταξύ. Αλλά το θέμα του προϋπολογισμού για τη ΣΜΚΙΟ είναι μόνο το 0,6% του προϋπολογισμού. Αυτό δεν είναι άλοθη για να δίδουμε χρηματοδότηση χωρίς ελέγχους. Αυτή είναι η πρώτη δήλωση. Δεύτερον, να διαλύσω την εντύπωση ότι εμείς λειτουργούμε σε πάρα πολύ δύσκολα και ε, επικίνδυνα θέατρα δεν ελέγχουμε, δεν αληθεύει αυτό. Όταν συνεργαζόμεθα με τις ΜΚΟ, το κάνουμε αφού έχουμε εξετάσει, αξιολογήσει τους εταίρους αυτούς. Αυτός είναι ένας βασικός δρόμος. Έχουμε 220 εταίρους, από τους οποίους 196 είναι ΜΚΟ. Εμείς ε, δεν δίνουμε κάθε χρόνο χρήματα σε όλες αυτές τις οργανώσεις. Έχουμε περιορισμού στον προϋπολογισμό μας. Δίνουμε σε 30% από όλες αυτές τις αιτήσια βάση χρήματα. Αλλά κάνουμε μια αξιολόγηση εξαντλητική και εξάντε, έτσι ώστε να δούμε αν τα κριτήρια γίνονται σεβαστά για τον κανονισμό μας, ε, μη ε, κερδοσκοπικές, πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μια χώρα μέλος ή στην χώρα στην οποία δίδουμε τα χρήματα και επίσης να συμμορφώνονται με κάποιες απαιτήσει οι οποίες δεν είναι μόνο χρηματοπιστωτικές αλλά και λειτουργικές. Δηλαδή ε, έγκαιρη παρέμβαση σε επίπεδα ανθρωπιστικών προβλημάτων, σε, σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών προβλημάτων. Έχουμε ένα ελεγκτικό περιβάλλον πολύ αυστηρό θα έλεγα και σε σχέση με την επιλογή αυτών που θα πάρουν χρήματα και μετά από την πρόταση για τον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος παρακολουθούμε πολύ ε, προσεκτικά τα χρήματα. Ένα από τα χαρακτηριστικά μας είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο τεχνικής βοήθειας. 450 άτομα τα οποία είναι επιτόπου εμπειρογνώμονες συνεργάζονται με τους εταίρους, συζητούν τα προβλήματα, παρακολουθούν και ελέγχουν. Και φυσικά, όπως και άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τους, τους ελέγχους εξ των υστέρων. Εκεί προσπαθούμε να δούμε και τι μπορούμε να διορθώσουμε από τις διαδικασίες που διαπιστώνει ότι δεν πήγαν καλά. Για 30 δευτερόλεπτα να μου επιτρέψετε να πω ότι το θέμα της διαφάνειας, να πω ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι υπέρ της διαφάνειας έτσι και αλλιώς. Η συζήτηση αυτή όμως μου θυμίζει κάποιες άλλες συζητήσεις, οι οποίες είχαν γίνει εδώ και 10 χρόνια, για το ποιοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι, αυτοί που ωφελούνται μάλλον τελικά. Ε, η αρχική οργάνωση, η επόμενη οργάνωση ή το σχολείο τελικά. Ή ε, η κυρία Α ή η κυρία Β η οποία ωφελείται από την χρηματοδότηση αυτή μετά από την παρακολούθηση σεμιναρίων κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι το επίπεδο λεπτομέρειας στο οποίο μπορούμε να φτάσουμε είναι δεδομένο. Η ΜΚΟ συνεργάζονται πολλές φορές ε, με τοπικές εκτελεστικές υπηρεσίες. Εμείς δεν έχουμε πολλές ε, σχέσεις με αυτές. Ε, τελικοί λοιπόν παραλήπτες των ποσών μας είναι η βασική μας συνεργαζόμενη εταίροι. Πριν από 10 χρόνια συμμετείχα στη συζήτηση για τα διαρθρωτικά ταμεία όταν μιλήσαμε για την διαφάνεια του τελικού δικαιούχου. Λέξη σιδηρόδρομο στα γερμανικά. Θέλαμε λοιπόν να υπάρχει διαφάνεια και σε επίπεδο κρατών μελών. Και μας ενδιαφέρει να δούμε σε ποιο βαθμό έχει ευοδοθεί αυτή. Εσείς ε, ε, μιλήσατε και για ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όπως ε, να μην είναι πολύ βαρύ και επαχθές το σύστημα ε, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο και στους συμπυρογνώμονες. Σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομο θα είμαι, διότι συμφωνώ με όσα είπε ο συνάδελφο και δεν υπάρχει λόγο να, να τα επαναλάβω. Θα αναφερθώ μονάχα σε ένα θέμα ε, όσον αφορά την εξωτερική ε, βοήθεια, αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτή είναι η μόνη εξάρτηση. Και επίση ε, το πώ ξέρουμε ότι οι οργανώσεις με τις οποίες ε, εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε είναι ανεξάρτητες, ε, κυρίως ε, όσον αφορά περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιοχές δηλαδή χώρες όπου η ελευθερία του συνεταιρίζεται, η ελευθεροτυπία ή η ελευθερία έκφρασης πολλές φορές δεν είναι αυτές που θα έπρεπε λόγω αυταρχικού περιβάλλοντος και στα πλαίσια του οποίου δύσκολα μπορούν, αν όχι αδύνατον είναι να εργαστούν ανεξάρτητα με κυβερνητικέ οργανώσεις. Πρέπει να σας πω ότι κατά αυτή την έννοια είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τα όσα κάνουν οι συνεργάτες μας προσπαθώντας να δημιουργήσουν ή να κρατήσουν ανοιχτό χώρο για συζήτηση και ε, ελευθερία λόγου. Ε, με μεγάλη προσοχή ακούω αυτά που λέγονται σχετικά με το ενδεχομένως κάποιο λόμπι να κρύβεται πίσω από κάποια ε, οντότητα. Δεν αντιλέγω και δεν αρνούμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ε, συμβαίνει. Ωστόσο, ε, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι θα πρέπει να βρούμε ε, μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις και τις υπόλοιπες πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες κάνουν καλή δουλειά αυτές οι οποίες αντιμετωπίζονται με εχθρότητα και από κυβερνήσεις και από, από συμφέροντα και παρόλα αυτά εξακολουθούν να εργάζονται σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να τα δούμε γιατί ε, αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να δουλέψουν και με τρόπο ανεξάρτητο ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την διευκρίνηση. Τώρα θα ζητήσω θα ζητήσω τον κύριο Άκερμαν να απαντήσει σε ερώτηση που του απευθύνθηκε. Ναι, νομίζω μία ερώτηση αφορούσε μας σχετικά ε, με την διαφάνεια Transparency International, ε, σχετικά με το αν έχουμε κάνει ε, κάποιες συγκριτικές μελέτες. Όχι. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μας απασχόλησε. Έχουμε όμως ε, κάποιες ε, ε, πληροφορίες σχετικά με την πρώτη μορφή της έκθεσης για την διαφάνεια και εμείς διευκρινίσαμε εκεί ότι τα ερωτήματα τα οποία εγείρονται σχετικά με την μη καταγραφή στο Μητρό διαφάνειας ε, αφορά πολλές ε, οργανώσεις. Ευχαριστώ λοιπόν για το κλείσιμο αυτό και τώρα πάμε ο δεύτερο μέρος. Πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή η αντίδραση από την πλευρά εκείνων που είναι και το θέμα προς συζήτηση. Καλέσαμε εκπροσώπους κάποιων οργανώσεων που θα λάβουν το λόγο. Βέβαια, δυστυχώς πρέπει να περιοριστούμε σε 5 με 6 λεπτά για τις αρχικές δηλώσεις. Μετά όμως θα λάβετε πάλι το λόγο στα πλαίσια της συζήτησης. Λοιπόν, ο κύριος Τόμας Χέκεμπερκ, ο πρώτος εκπρόσωπος ΜΚΟ, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκπαίδευσης Κατάρτισης και μέλος του τη Civil Society Europe. Ε, ε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίπερ, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Ως πρώτος ομιλητής μιας οργάνωσης από την κοινωνία των πολιτών θα πω ορισμένα βασικά. Δηλαδή, γιατί χρηματοδοτούμε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τι ρόλο παίζουν αυτές στην κοινωνία μας είναι σημαντικό κομμάτι της πλουραλιστικής δημοκρατίας και προσφέρουν πολλές υπηρεσίες ευραίως φάσματος. Εκπροσωπούν, και αυτό είναι σημαντικό, την ευρωπαϊκή ε, κοινωνία και τα διαφορετικά συμφέροντα των πολιτών και τα ενδιαφέροντά τους. Και για να απαντήσω σε μια ερώτηση, ο κύριος που έκανε ερώτηση δεν είναι εδώ. Γιατί έρχονται στο γραφείο του εκπρόσωποι των ΜΚΟ και τους στέλνουν ε, mails γιατί εκπροσωπούν ένα ευρύτερο κύκλο ανθρώπων, όχι για ίδιο συμφέρον, παρόλο που αυτό πολλές φορές δεν εντάσσεται μέσα στη λειτουργία του πολιτεύματος ε, ή το, της πολιτικής. Όμως ε, λειτουργεί στα πλαίσια ενός πολιτεύματος που στηρίζει και άλλους. Η η δημόσια χρηματοδότηση των ΜΚΟ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε μια πλουραλιστική ανοιχτή κοινωνία ε, είναι απαραίτητη. Τονίζω εδώ τη δημόσια χρηματοδότηση. Αυτό δεν σημαίνει, όπως ακούστηκε κανένα δυο φορές εδώ, ότι οι οργανώσεις αυτές παίρνουν χρήματα από την κυβέρνηση. Όχι. Δεν παίρνουν τα χρήματα της κυβέρνησης, παίρνουν από το κράτος ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα για τον απλούστατο λόγο ότι εκπροσωπούν ένα κομμάτι της κοινωνίας, δηλαδή ένα κομμάτι ε, ε, που θέλει να είναι εξάρτητο από τις κυβερνήσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενώ είναι κομμάτι του κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάποιες κυβερνήσεις που μόλις ανέλαβαν το πιδάλιο ε, περιόρισαν πολύ τον πλουραλισμό στη χώρα τους ε, και αυτό εκδηλώθηκε μεταξύ άλλων από την πάυση της χρηματοδότησης ΜΚΙΟ. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει έναν ακόμα σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση ΜΚΙΟ γιατί σε ορισμένες χώρες οι οργανώσεις αυτές δυστυχώς ε, αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα λόγω της κυβερνητικής αυθαιρεσίας. Πρέπει να πω όμως παράλληλα ότι πιστεύουμε ότι οι οργανώσεις όπως και αν αυτές ονομάζονται που ε, τάσσονται κατά των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολεμούν βεβαίως και δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να υποθεί ξεκάθαρα. Σχεδόν όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στον ορισμό των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι δύσκολος ο ορισμός ας πούμε, μη κοιό σημαίνουν ακριβώς αυτό, δηλαδή θέλουν δημόσιο χρήμα, κρατικό χρήμα όχι ε, κυβερνητικό χρήμα, αναφέρθηκε το πολωνικό παράδειγμα που είναι μπερδεμένο και δεν ξέρουν εκεί ποιος ακριβώς κρύβεται πίσω από ε, τις ΣΜΚΙΟ. Εμείς από τη δική μας τη Σκοπιά πιστεύουμε ότι πρέπει ίσως να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα να βρούμε έναν καλό ορισμό για τις ΜΚΟ ή για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή να βρούμε έναν άλλον ορισμό. Ίσως θα πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια ακόμη. Πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εδώ και 30 χρόνια προσπαθούν να βρουν μια λύση και σήμερα ε, ε, ελέγχθη ότι ναι, είναι πολύ δύσκολο γιατί έχουμε 28 διαφορετικές λύσεις σε κάθε κράτος μέλος. Υποθέτω ότι το 70% των νόμων που περνούν από εδώ δεν διαφοροποιούνται 28 φορές. Γιατί λοιπόν να μην προσπαθήσουμε να βρούμε και έναν ορισμό ενίο για τις ΜΚΟ. Η επίσημη δήλωση της Κομισιόν μέχρι τώρα είναι ότι δεν υποβάλλουμε πρόταση γιατί δεν πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή θα περάσει από το Συμβούλιο. Αν το είχαμε αν, αν, αν σκεφτόμαστε όλοι έτσι, τότε οι επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα ξεπερνούσαν τις πέντε σελίδες. Πιστεύομαι λοιπόν ότι είναι ευκταία αυτή η προσπάθεια εξέβρεσης ορισμού για τις ΜΚΟ και τις παρεμφερείς οργανώσεις. Τέλος, και δεν θα μακρηγορήσω πάνω σε αυτό, ε, η ορατότητα, visibility της χρηματοδότησης. Αναφέρθηκε εδώ από τους ε, εμπειρογνώμονες ότι ε, δεν τηρούνται οι προδιαγραφές. Οι περισσότερες ΜΚΟ τηρούν τις προδιαγραφές που τους δίνει η εκτελεστική εξουσία ή η ε, Κομισιόν. Σίγουρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτιώσεις. Μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα τα πράγματα, κάνουμε την αυτοκριτική μας, αλλά θα ήταν μια μεγάλη ανακούφιση για μας αν υπήρχαν ενιαίες διατάξεις και προδιαγραφές από την Κομισιόν ώστε να μην διαφοροποιεί κάθε γενική διεύθυνση τις ε, προδιαγραφές της. Αυτό θα ε, απλούστευε πολύ τη δουλειά μας. Εδώ δεν πρόκειται, ε, πρόκειται και για δημοσιεύσεις, όχι μόνο για σελίδες στο διαδίκτυο. Ε, σίγουρα ε, η ορατότητα δεν γίνεται με ε, τρόπους ε, εντυπωσιακούς και αλλά με τρόπο συστηματικό. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί θα πρέπει να προεστιάσουμε τις προσπάθειες. Αυτά για τις ΜΚΟ, το ρόλο τους, τη χρηματοδότηση, την προσπάθεια εξέβρεσης ορισμού και τη βελτίωση της ορατότητας των, των κονδυλίων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ για τα επιχειρήματα που προβάλλατε. Τώρα, ε, η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Κάτριν Σίκα από μια εθελοντική οργάνωση συνεργασίας σε κατεπίγουσες καταστάσεις. Εγώ θα μιλήσω αγγλικά παρότι θα μπορούσα να εκφραστώ και στη γερμανική. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τον τρόπο με τον οποίο ε, υλοποιούν την ε, δράση, της, ε, τη δράση τους. Προηγουμένως ακούστηκε από πλευρά της Κομισιόνη γιατί ε, συνεργάζεται με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όσον αφορά την, τις ανθρωπιστικές επίγουσες καταστάσεις, η εκρίζωση της φτώχεια και η αντιμετωπίση επίγουσων καταστάσεων είναι ο κύριος στόχος. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα της ε, Κομισιόν ε, που επιβεβαιώνουν ότι χρειάζον, χρειάζεται η Κομισιόν την, της εμικιό έτσι ώστε να υλοποιήσει η Κομισιόν τα προγράμματά της ΜΚΟ οι οποίες έχουν την ικανότητα βέβαια να υλοποιήσουν προγράμματα. Πολλοί λόγος γίνεται εδώ για την Κομισιόν, αλλά ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και ε, τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις, έστω και αν κάποιες διαδικασίες μπορεί να είναι αμφισβητούμενε, α πούμε, από αυτές που εφαρμόζονται σε κάποιες χώρες μέλη. επανειλημμένα έχει αποδεχθεί ο ρόλος και η σημασία ε, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την ενδυνάμωση και ε, εφαρμογή της ε, δημοκρατίας. Υπάρχουν πολλά συγκριτικά πλέον εκτήματα στη συνεργασία με τις ΜΚΟ και αυτό το έχουν αναγνωρίσει επανειλημμένα και ο Ερυθρός Σταυρός και τα Ηνωμένα Έθνη. Στην ουσία, λοιπόν, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει βρίσκονται επί τόπου ε, με τρόπο που δεν μπορούν και με παρουσία που δεν μπορεί να αντικατασταθεί ε, από άλλου. Ε, Στι πήγουσε ανθρωπιστικέ καταστάσει, οι ΜΚΟ είναι αυτέ οι οποίε και στη, στο Χαλέπι και στη Σομαλία και στην Ιγυρία βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή έτσι ώστε να προωθήσουν και να μοιράσουν την ανθρωπιστική βοήθεια και με τον τρόπο αυτό βοηθούν την μακροπρόθεσμη ε, ανάπτυξη την οποία ε, επιδιώκεται σε αυτές τις ε, χώρες. Γιατί οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν την δυνατότητα να εργαστούν με τρόπο διαρκή και βιώσιμο. Ε, επίσης, οι ΜΚΟ έχουν προστιθέμενη αξία ε, λόγω του ότι έχουν την δυνατότητα γρήγορα να προσαρμοστούν σε καταστάσεις οι οποίες με ταχύ ρυθμό ε, αλλάζουν κυρίως σε περιπτώσεις συγκρούσεων ή ευάλωτων χωρών. Επίσης, οι ΜΚΟ είναι αυτές οι οποίες μπορούν να δουλέψουν με αποτελεσματικότητα, επαγγελματισμό και γνώσεις και μάλιστα πριν ε, δώσει χρήματα η Κομισιόν και πριν κάνει η Κομισιόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρήσουν ε, ε, το ενδεχόμενο συνεργασίας με αυτές τις ΜΚΟ. Αυτοί οι εταίροι βρίσκονται ήδη επιτόπου ε, και ε, εάν μετά από δύο-τρία χρόνια δεν έχουν την δυνατότητα ε, να παραδώσουν αποτελεσματικό έργο, βγαίνουν από την εικόνα. Με ενδιαφέρον ιδιαίτερο άκουσα εδώ τον συνάδελφο από το ελεγκτικό συνέδριο να αναφέρεται στον κατακαιρματισμό των χρηματοδοτήσεων και των projects. Ναι, μα γι' αυτο ακριβω ακριβώς υπάρχουν δύο-τρει μεγάλε οργανώσει, οι οποίε παίρνουν τα περισσότερα χρήματα γιατί έχουν την δυνατότητα να προωθήσουν ε, ε, ε, πολλά προγράμματα. Τώρα, εάν έτσι θα πρέπει να συνεχιστεί ή αν κοινωνικά έτσι θα πρέπει να, η κοινωνία έτσι θα πρέπει να προχωρήσει, δηλαδή με μεγάλους θεσμοθετημένους οργανισμούς και μικιό, αυτό δεν το ξέρω. Πάντως, σε ολόκληρη την Ευρώπη, εσείς που εκπροσωπείτε όλες τις χώρες και όλες ε, τις περιοχές ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω ότι κατανοείται ότι επιτόπου οι ανάγκες είναι πολλές και περίπλοκες και επομένως χρειάζονται operators οι οποίοι να γνωρίζουν το πώς να κινηθούν επιτόπου. Επίσης, όταν μιλάμε για ανθρωπιστική βοήθεια, υπάρχει ισχυρή δέσμευση ε, συνεργασίας με τους τοπικούς ε, ε, φορείς που η Κομισιόν δεν το επιτρέπει για την ώρα. Εμείς πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματα θα δαπανηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο έχει υποβληθεί στην Κομισιόν. Επίσης, ε, σε, ε, αναρωτιέμαι αυτά που ακούγονται σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αναρωτιέμαι γιατί, γιατί ε, ε, υπάρχει τέτοια πίεση γιατί και εγώ πληρώνω φόρους και η οικογένειά μου πληρώνει φόρους. Εάν ε, προκύπτει ας πούμε ένα σκάνδαλο σε μία ε, ε, τότε γίνεται μεγάλη συζήτηση. Όχι όταν κάνουν τα πολλά καλά, όταν κάνουν το ένα ε, λάθος. Και ξέρετε, όλοι υφιστάμεθα ε, πιέσεις και επομένως όλοι σε κάποια περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά και επομένως όλοι θέλουμε να λειτουργήσουν τα πράγματα καλά και βάσει της... Και εδώ λίγο ε, αμφισβητώ την έννοια της απόλυτης αναλογικότητας στο δικό μας τομέα. Ο Σάνθος εδώ έδωσε πολλά στοιχεία και από τη στιγμή που αναφέρονται επανειλημμένα τα διαφορετικά ταμεία θα ήθελα να πω ότι το εκτιμούμενο ποσοστό λάθους είναι 2,8 100% ε, ε, την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου του 2015 που είναι το, η τελευταία δημοσιευμένη έκθεση. Ε, και και 5,2% ε, είναι το, περι, το περιθώριο λάθους για τα διορθωτικά προγράμματα εδαφικής συνοχής κτλ. Ε, και ε, η Global Europe ας πούμε έχει ένα συνολικό ποσοστό λάθους 4% ε, ενώ τα διευθυντικά ταμεία μπορεί να φτάνουν και στο 51%. Να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως είναι ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αλλά κάθε οργάνωση η οποία δέχεται χρηματοδότηση ή επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει για κάθε πρόγραμμα ε, να υποβάλει όλα τα σχετικά ε, δικαιολογητικά. Ε, ε, είναι πολλοί οι ε, δωρητές και επομένως υπάρχουν περιπτώσεις όπου η μη κυβερνητική οργάνωση θα πρέπει να υποβάλει εκθέσεις σε κάθε ένα ξεχωριστά δωρητή. Σε γενικές γραμμές πάντως και συμπεράσματι μπορώ να πω ότι η πλευρά των μη κυβερνητικών οργανώσεων δέχεται τις προτάσεις όσον αφορά τις νέες προτάσεις συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και βεβαίως αποδέχονται και τις αρχές για εσωτερικό και εξωτερικό οικονομικό έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Σίκ για όσα μας σας είπατε. Εμείς είμαστε στο πλευρό σας, μην νομίζετε ότι πρέπει να υπερασπίσετε τη θέση σας, αλλά παρόλα αυτά ε, ακούσαμε πολύ προσεκτικά και θετικά. Πρώτο ο ομιλητής, ο κύριος Σίμους Τζέφερσον, ο οποίος είναι διευθυντής της Ομοσπονδίας Ανακούφισης και Ανάπτυξης. Ε, ναι, έχετε το λόγο. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Ένα είναι το θέμα το οποίο τονίζει ιδιαίτερα η έκθεση αυτή και έχει ε, σχέση με την λειτουργία των ΜΚΟ μεταξύ τους σε συνεργασία, σε επίπεδο συμμαχιών. Ίσως να υπάρχουν κάποιες παρανομήσεις για τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό και για τα κίνητρα τα οποία θα μπορούσαν ε, να μην έχουν ε, ξεκάθαρους στόχους. Λοιπόν, να σας εξηγήσω γιατί συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Καταρχάς, όταν εργάζεται κανείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει σημασία το να συνεργαζόμαστε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήγουμε σε εκείνες θέσεις και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλο. Νομίζω ότι όλα τα μέλη, και εγώ προέρχομαι από μια συγκεκριμένη συνομοσπονδία, και όλα τα μέλη της συνομοσπονδίας ωφελούνται από τη στενή συνεργασία μεταξύ των ΜΚΟ από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Το δεύτερο είναι οι οικονομίες κλίμακας και ο τρόπος με τον οποίο καταλήγουμε σε συνενέσεις πάνω σε θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα υπάρχει και αν θέλετε μία έννοια αλληλεγγύη στον τομέα μας. Έχουμε μικρές και μεγάλες και νομίζω ότι ακριβώς ένα τμήμα αυτής της προσπάθειας τεκμηριώνεται από τη δράση μας. Ε, οι συμμαχίες αυτές βοηθούν και τους συνομιλητές μας και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις συμμαχίες αυτές και τις συνομοσπονδίες. Γιατί μερικές φορές ε, περίπλοκες και διαφοροποιημένες μεταξύ τους προτάσεις εμείς τις συγκεντρώνουμε ε, και στην αναζήτηση της ε, παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας ο τρόπος που το κάνουμε αυτό είναι καλύτερος από ό,τι αν γίνονταν μεμονωμένα. Πολλά από τα μέλη της δικής μου ε, συνομοσπονδίας ανήκουν και σε άλλα δίκτυα. Δεν είναι κάτι το αρνητικό αυτό. Νομίζω ότι σε διάφορους τομείς συμβαίνουν αυτού του είδους τα φαινόμενα Υπάρχουν ΜΚΟ που εργάζονται και στον τομέα τον ανθρωπιστικό, σαν παραδείγμα το δίκτυο Voice της παρακαθημένης μου σε θέματα που ασχολούνται με παιδιά, σε τομεί συγγνώμη που ασχολούνται με τα παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα το ασυνήθιστο δηλαδή, αν μία οργάνωση ανήκει σε διαφορετικά δίκτυα βλέπουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο αρκετά συχνά. Ο τρόπος με τον οποίο δίδονται τα θύματα στα δίκτυα, τα χρήματα στα δίκτυα, είναι κάτι το οποίο έχει ε, αντιμετωπιστεί από τους προηγούμενους ομιλητές. Ε, βλέπουμε εμείς ότι και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ο έλεγχος ο οποίος μας γίνεται ο λογιστικός είναι πάρα πολύ ισχυρός. Δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο σε σχέση δηλαδή με το τι ακριβώς κάνουμε. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την διαφάνεια ε, προς όφελος του φορολογούμενου. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα της λειτουργίας σε επίπεδο συμμαχιών είναι κάτι το οποίο βοηθά τα μέλη μας, βοηθά τις ΜΚΟ και ε, θα βοηθήσει και βοηθά επίσης ε, και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και όλους τους εμπλεκομένους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναδείξατε το ρόλο των δικτύων. Σίγουρα θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Ε, σε σχέση με την ανάγκη τεκμηρίωσης ε, κάποιων χρηματικών ροών. Γιατί ε, σίγουρα δημιουργούνται συνέργειες, αλλά ίσως κάποια επιμέρους μπορεί να διαμορφώνονται με διαφανέστερο τρόπο. Τέλος, πολύ σημαντικός, ο κύριος Τζέρεμι Βέιτς, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Γραφείου, μέλος του Green 10. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω στη συζήτηση αυτή. Είμαστε πεπισμένοι στις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Ε, σαφώς είμαστε υπέρ της ενίσχυσής τους. Ε, κυρία, είπατε, απαντώντας στην κυρία Σίκο, ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά την ουσία της δουλειάς μας και τη στηρίζετε. Οπότε αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε εδώ είναι ότι η χρηματοδότηση από την Κομισιόν στις ΜΚΟ συμβάλλει πολύ σημαντικά στην αποτελεσματικότητά μας. Πρέπει να πω ότι είναι δύσκολο, θεωρώ, να αναγνωρίσω τη δουλειά που κάνω ως ε, γενικός γραμματέας στη μεγαλύτερη περιβαλλοντική οργάνωση. Είναι δύσκολο να καταλάβω ορισμένε παρατηρήσει που ακούστηκαν, τώρα έφυγαν οι κύριοι, γιατί η δική μας εμπειρία είναι ότι ε, οι ε, αιτήσει που δεχόμαστε είναι λεπτομερέστατες και οι διαδικασίες είναι λεπτομερείς, με λεπτομέρειες για όλα τα θέματα γιατί αναφέρθηκε ότι σε κάποια θέματα υπάρχει έλλειψη διαφάνειας. Πραγματικά εκπλήσωμαι ακούγοντας τέτοιες δηλώσεις στην αίθουσα αυτή. Η προοπτική που προβάλλω εδώ ε, ε, επιβεβαιώνεται αν θέλετε και από την έκθεση που έγινε γιατί η EB ε, επελέγει ως μία μελέτη περίπτωσης εμείς είμαστε πολύ ανοιχτοί στη μάθηση, θέλουμε να γινόμαστε ακόμα πιο διαφανείς. Αλλά σε σχέση με την EB, τα ε, αποτελέσματα ήταν καλά στην έκθεση. Πολλά κάνουμε σωστά. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα καλύτερα. Ε, στη, για να δείτε τα μέλη, τα βλέπετε με αλφαβητική σειρά κατεβαίνω κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Ε, αλλά αν μόνο αυτή είναι η κριτική, ότι δηλαδή παίρνει χρόνο για να τα δούμε όλα τα μέλη, ε, αυτό σημαίνει ότι πολλά κάνουμε καλά. Ε, έχω γράψει ορισμένα βασικά ε, το, η τρίτη και η τέταρτη παύλα είναι σημαντικές γιατί αναδεικνύουν τη σημασία της χρηματοδότησης των ΜΚΟ. Διότι αν αφαιρεθεί η χρηματοδότηση αυτή από τις ΜΚΟ, τότε θα δημιουργηθεί μεγάλη έλλειψη ισορροπίας και οι εμπλεκόμενοι δεν θα μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά. Οι εμπλεκόμενοι μέσω των ΜΚΟ μπορούν να προσέρχονται ε, σε τράπεζες συζητήσεων μαζί με τους ε, ενδιαφερόμενους από τον ιδιωτικό τομέα και έτσι η διαδικασία λήψης αποφάσεων γίνεται με πιο ισόρροπο τρόπο. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ε, σύμβαση του Άρχους, αλλά και με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την νομική υποχρέωση όχι να τις χρηματοδοτεί, αλλά να στηρίζει τις ΜΚΟ σε πολλούς τομείς και διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Και ε, όλα αυτά θα ήταν πολύ ακαδημαϊκά αν δεν συνοδεύονταν και από απτή υποστήριξη, οικονομική δηλαδή. Έχω και προσωπική εμπειρία, ένα παράδειγμα. Όταν οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονταν τη πρότυπα για τις εκπομπές ε, ρήπων Εκεί είναι ένας τριμερής διάλογος, ε, γίνεται δηλαδή και με την κοινωνία των πολιτών και με τις επιχειρήσεις ε, ο διάλογος, αλλά η κοινωνία των πολιτών εκπροσωπείται από λίγες μονομίκιο, ακριβώς γιατί προβλέπεται δημόσια χρηματοδότηση. Ε, κάποιοι θα ήθελαν να γίνεται ο διάλογος μόνο μεταξύ κυβερνήσεων και ε, βιομηχανίας ή επιμέρους κλάδων. Ε, δεν το θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε τέτοια κοινωνία. Και δυσκολεύονται τα πράγματα ακόμη περισσότερο όταν ε, πολλά κυβερνητικά στελέχη είναι εκπρόσωποι των κλάδων της βιομηχανίας. Μην ξεχνάτε το σκάνδαλο Dieselgate που ήταν ξεκάθαρο παράδειγμα που έδειχνε δηλαδή ότι ε, ο ιδιωτικός τομέας και οι κυβερνήσεις ε, συνεργάζονταν υπερβολικά στενά, ενώ η ΜΚΟ μπορεί να επηρεάσουν ε, θετικά πολλά θέματα, όπως θα μπορούσαν δηλαδή να είχαν προλάβει και το σκάνδαλο, παίζοντας πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις εκπομπές. Ε, μου φαίνεται πρέπει να κλείνω σιγά σιγά. Ε, να πω τέλος ότι είμαστε υπέρ ενός μητρώου διαφάνειας υποχρεωτικό που θα δημοσιεύει τα ονόματα όλων των ομάδων συμφερόντων. Ε, έτσι θα διαφοροποιηθούμε από τους λόμπις. Και θέλουμε περισσότερη ε, υποχρεωτική ε, νομοθεσία για αυτό το σύστημα. Ε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και ένα φιλικό προς το χρήστη και συνεπές ε, δημοσιονομικό σύστημα διαφάνειας. Σταματώ εδώ για να αφήσουμε χρόνο και στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Όλοι οι πολιτικοί ανεξάρτητα κόμματος Όλοι οι πολιτικοί ωφελούμεθα από τη δουλειά σας και γι' αυτό την εκτιμούμε τη δουλειά σας. Βεβαίως ε, πρέπει να τεκμηριώνεται η δουλειά αυτή. Δεν θα πρέπει να στηρίζεται σε μύθους και προκαταλήψεις. Ε, χρειάζονται κριτήρια για την υποστήριξη. Μπορούν να προσθεθούν αυτά. Και προφανώς η κριτική, αυτό το ξεκαθαρίζω όλο και περισσότερο, δεν απευθύνεται στις ΜΚΟ, πρόκειται για την εμπιστοσύνη. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή, ε, θα έπρεπε τα νούμερα, τα στοιχεία, τα αριθμητικά να παρουσιάζονται με πιο καλό τρόπο. και σε αυτό το ζήτημα μπορεί να παίξει μεγαλύτερο ρόλο το ελεγκτικό συνέδριο που θα μας δώσει τα στοιχεία εκείνα που θα μας βοηθήσουν να οικοδομηθεί ε, εμπιστοσύνη. Λοιπόν, το επίσημο πρόγραμμα τελείωσε. Δύο ε, ε ζήτησαν το λόγο, δύο συμμετέχοντες. Α, τρίτος ε, ο συνάδελφος Στάς και θα πρέπει να τελειώσουμε στις 6.30 το αργότερο γιατί ακολουθεί και άλλη εκδήλωση. Λάουρα Ντασίλβα από τη ΜΚΟ Monitor. Πού είναι? Α, μάλιστα. Στα πίσω καθίσματα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω που φέρατε το θέμα αυτό σε συζήτηση. Να αναφέρω ότι η έρευνά μας συγκεντρώνεται στο θέμα της χρηματοδότησης της Ένωσης ε, προς περιοχές και χώρες εκτός της Ένωσης. Έχουμε καταλήξει σε πολλά κοινά συμπεράσματα με τα δικά σας Πολλές από τις συστάσεις σας είναι συστάσεις τις οποίες συμμεριζόμεθα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στον κόσμο με 18 με 82 συγγνώμη δις ευρώ. Ένα τμήμα αυτών των χρημάτων πηγαίνουν στις Σμικιώ. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το ποσό βέβαια που καταλήγει στη ΜΚΟ. Δυστυχώς το σύστημα δεν είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς πόσα χρήματα πηγαίνουν στη ΜΚΟ. Το 100% αφορά θέματα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ΔΕΦΚΟ και της ΕΚΟ τα δεδομένα αυτά δεν τα, δεν έχουμε εμείς επεξεργαστεί και είναι σημαντικό να ξέρουμε το τι γίνεται εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν διαρωτώμε τι μπορούμε να κάνουμε για την καταμέτρηση των επιπτώσεων της παρέμβασής μας μέχρι σήμερα το θέμα δεν είναι μόνο θέμα διαφάνειας. Μια οργάνωση που παίρνει χρήματα πιστεύει ότι κάνει καλά ορισμένα πράγματα αλλά να μην ικανοποιεί πλήρως τις επιθυμίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση επί τόπου και επίσης και ο διάλογος με τις ΜΚΟ από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσε να υπάρξει ένας διάλογος ο οποίος να λαμβάνεται υπόψη τους τοπικούς εταίρους. Και αναφέρομαι και σε ΜΚΟ που δεν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρηματοδοτεί προγράμματα που θεωρεί κατάλληλα, αλλά τελικά όμως ε, οι μοικείο που παίρνουν τα χρήματα αυτά κατηγορούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κακή διαχείριση. Ευχαριστούμε για τα επιχειρήματά σας. Η κυρία Κόνι Ρόιτερ από την Σολίντα. Oh, α, συγγνώμη. Κόνι, Κόνι είναι ανδρικό όνομα. Α, για την αδερφή μου Κόνι τη λένε, λέει ο πρόεδρος. Είμαι Γενικός Γραμματέας της Solidar που είναι Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Είπατε πριν ότι είναι δύσκολος ο ορισμός της ΜΚΟ. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν οργανώσεις μέλη. Έχουμε την Κάρτα στη Ολιντάρ, στη Γερμανία έχουμε την ε, ε, οργάνωση ε, που βοηθάει τους εργαζομένους. στα δίκτυά μας, ε, μια φορά που μετρήσαμε, συμπεριλάβαμε 9 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό που είναι λίγο λυπηρό είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη υπάρχει ε, ένα άρθρο 11 που αφορά την χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση των ΜΚΟ κοινωνικών δικτύων έχει να κάνει με το πώς επικοινωνούν τα θεσμικά όργανα της Ευρω... Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών. Ε, υπάρχει ε, μια ε, αμέλεια εδώ, διότι δεν τονίζεται επαρκώς η διαφάνεια αλλά και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Επίσης είναι κρίμα που οι συνάδελφοι ε, προέβαλαν σωστά πολιτικά επιχειρήματα, αλλά πρέπει παράλληλα να δούμε και τη νομική μας κάλυψη. Ένα ευρωπαϊκό δίκτυο θα πρέπει να πάει στο συμβολογράφο, θα πρέπει να ε, ακολουθεί ε, το, ε, την νομοθεσία κάθε χώρας. Δηλαδή, σε κάθε βήμα ε, με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ακολουθείται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, τέλος, θα είμαι θα ευγνώμονε στο Κοινοβούλιο αν η Επιτροπή σας υπογράμμιζε πόσο σημαντικό είναι ε, ένα ευρωπαϊκό καθεστώς για τις ΜΚΟ, διότι έτσι θα διασφαλίζεται το πλήρης διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ε, ενιαία ε, πρότυπα και διαδικασίες. Αυτό το θέλουμε όλοι. Ε, και έχουμε έναν ομιλητή ακόμη, τον συνάδελφο Στάις. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι θεωρώ την ακρόαση αυτή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούσαμε ε, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και από εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων και ε, άλλους. Πρέπει να πω ότι το θέμα παρουσιάζεται με αρνητικό πρόσημο πολύ συχνά. Ωστόσο, τα πράγματα λειτουργούν και λειτουργούν καλά, ακόμα και με λίγα χρήματα, ακόμα και με κατακαιρματισμό κτλ. Κοιτάξτε, και τα πολιτικά κόμματα ε, και διάφορα ε, ιδρύματα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούνται από δημόσιο χρήμα. Πρέπει να τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Και νομίζω ότι ε, είναι πολύ ε, σημαντικό ε, να καταλάβουμε ότι τέτοιου είδους εκπρόσωποι ας πούμε και μη κυβερνητικών οργανώσεων δίνουν λίγο φρέσκο αέρα στους τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ακούμε προσεκτικά ε, αυτά που μας λένε και γι' αυτό είναι σημαντικό να εξακολουθήσει να υπάρξει ε, αυτή η διασύνδεση. Ε, στην σελίδα 98 της μελέτης ε, γίνεται λόγος για ορατότητα. Ε, εγώ νομίζω ότι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, είναι θεμητό να γίνεται τέτοια αναφορά στην ορατότητα ναι, και θα πρέπει οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ να αναφερθούν στο θέμα αυτό. Ε, ε, ζητώ συγγνώμη, εγώ σε τρία λεπτά θα πρέπει να φύγω ε, γιατί πρέπει να είμαι αλλού, αλλά ελπίζω κάποιο να μου μεταφέρει την απάντηση. Σε τρία λεπτά θα έχουμε τελειώσει. Η κυρία Σίκ θα απαντήσει από τις ΜΚΟ. Θα ξεκινήσω εγώ και μετά μπορεί να προσθέσουν κάτι οι συνάδελφοι. Να πω ότι έχουμε δουλέψει ε, πολύ με την Επιτροπή Ίντε και νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε και πώς μπορεί η συνεργασία μας ε, να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Ε, είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε κάθε νομική πτυχή της ορατότητας. Αλλά βεβαίως σίγουρα ε, πρέπει να υπάρχει ορατότητα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωση, ε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η απαραίτητη διασύνδεση ανάμεσα στην ενωσιακή και τις εθνικές πολιτικές. Εννέα στους 10 Ευρωπαίους πολίτες υποστηρίζουν την αναπτυξιακή και ανθρωπιστική, ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι έχει ε, αυξηθεί το ποσοστό αυτό σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο και εάν η αποδοχή είναι τόσο ψηλή, αυτό σημαίνει ότι ε, κάτι κάνουμε καλά. Ja. Bitte, noch ein. Thank you. Perhaps uh, a, a last point from me, and it's to do with. Και εγώ να πω κάτι τελευταίο σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα, εκ, αντι, αντιπροσωπευτικότητα. Εμείς προσπαθούμε πραγματικά να είμαστε αντιπροσωπευτικοί και ακριβώς ε, για, για λόγους ε, δημοκρατικής λογοδοσίας ε, προσπαθούμε όντως να είμαστε υπόλογοι απέναντι στους δωρητές μας και απέναντι στους υποστηρικτές μας και φυσικά δίνουμε λογαριασμό και σε όσους μας υποστηρίζουν και που παρακολουθούν προσεκτικά το έργο μας. Ε, αναφέρθηκαν οι αρχές ε, της ε, Κωνσταντινούπολης, Istanbul Principles, αναφέρθηκαν και άλλες αρχές. Εμείς ως οργανώσεις θεωρούμε ότι πρέπει να δίνουμε λόγο και στους εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες που μας στηρίζουν και εξ ονόματος των οποίων δρούμε. Επίσης, ε, δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να δίνουμε λογαριασμό μόνο για τα οικονομικά, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους, όλες τις υπόλοιπες ε, ε, πλευρές της δράσης μας. Πρέπει να δίνουμε λογαριασμό όντως, γιατί χρησιμοποιούμε χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμμετασχόντες ε, μάθαμε πράγματα σήμερα. Ε, ευχαριστώ πολύ και για τον πειθαρχημένο τρόπο της διεξαγωγής της ε, συνάντησης αυτού του workshop. Θα δούμε τώρα τι συνέχεια θα πάρει η έκθεση. Προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας. Εξ ονόματος κυρίας Γκρέσλε επίσης ε, να σας δώσω πολλούς χαιρετισμούς.